Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη συνεδρία της, της συνεδρίασής μας εσωτερικής... της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Θα ήθελα πολύ θερμά να καλωσορίσω τον Επίτροπο Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την εσωτερική αγορά και θα θέλω να τον ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερω γιατί ήταν και χθε το απόγευμα. Και χθε το απόγευμα και σήμερα το πρωί 9 η ώρα ακριβώς χωρίς να καθυστερήσει καθόλου. Ήταν μάλιστα εδώ και πριν έρθουν τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλα τα μέλη της ομάδας σας. Είναι πολύ γνωστά πρόσωπα που ε, βρίσκονται στα έδρανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και καλύπτουν διάφορες πτυχές εργασίας σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς ε, και την ομάδα σας γιατί είστε πάρα πολύ διαθέσιμοι και μιλώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων. Πραγματικά εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος την συνεργασία με την ομάδα σας. Είναι πάντοτε διαθέσιμοι να απαντούν στα ερωτήματά μας, να μας δίνουν νέες ιδέες, να αναλαμβάνουν νέες πρωτοβουλίες και έχουμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία μαζί τους. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει αυτό. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και στοχευμένο διάλογο σήμερα με τον Επίτροπο. Αφορά το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας για το 2010-2011 ενημερώθηκα ότι 30% του προγράμματος θα μας ε, αναφέρεται σήμερα. Είναι, όχι μόνο, είστε μόνο, όχι μόνο ένα, ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά έχετε και πολλή δουλειά να κάνετε. Μου ζήτησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, να καλέσω όλους τους ε, αρμόδιους ε, υπουργού, ε, συγγνώμη, επιτρόπους να μας υποβάλουν το πρόγραμμά τους και θα συζητηθεί αυτό στην διάσκεψη των προέδρων. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω στο πρώτο, στον πρώτο γύρο συζήτησης να επικεντρωθείτε περισσότερο στα ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα εργασίας για την εσωτερική αγορά. Μέχρι τις 10 και 4 θα είναι μαζί μας ο Επίτροπος. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός για ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα εργασίας, γιατί αυτό, αυτός είναι ο στόχος μας σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε. Η Γραμματεία έχει ετοιμάσει μία σύνοψη για να μπορέσετε να ε, διαβάσετε καλύτερα αυτό το πολύ μακροσκελές έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθήσαμε να, να χρησιμοποιήσουμε έναν φιλικό προς το χρήστη ε, τρόπο παρουσίασης των προτάσεων ε, για να μπορείτε να εντοπίσετε τις προτάσεις που ενδιαφέρουν περισσότερο την Επιτροπή μας. Είμαι σίγουρος ότι ο Επίτροπος θα σας αναφέρει πολύ περισσότερα. Σας δίνω την δυνατότητα να λάβετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεν χρειάζεται να σας ξαναπώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι εδώ, γιατί έχω πάρα πολύ καλές αναμνήσεις. Δεν κάνουμε πολιτική με την νοσταλγία, πρέπει να έχουμε καλά, καλές αναμνήσεις. Και εγώ έχω καλές αναμνήσεις από την Επιτροπή σας. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους μου από τη Γενική Διεύθυνση Αγορών που είναι εδώ. Ε, να τους ευχαριστήσω για την διαθεσιμότητά τους και τη βοήθειά τους και θα ήθελα να ε, ακούσω την άποψή σας για το πρόγραμμα εργασίας μου. Η Κριστίν Ορλά είναι εδώ μαζί μου που είναι υπεύθυνη της ομάδας μου και ο υπεύθυνο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι επίσης μαζί μου. Πρόκειται για ερωτήματα που με έχουν απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ και 60 χρόνια η ΕΚΑΧ, ε, ο πρώτος λίθος ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετήθηκε, μετά είχαμε την κοινή πολιτική, μετά την ενιαία αγορά. Τι περιμένουν σήμερα οι πολίτες μετά από 60 χρόνια που έγινε το πρώτο βήμα οι περισσότεροι, κάποιοι λένε «Ε, δεν περιμένουμε και πάρα πολλά. Εγώ νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Νομίζω ότι ο καταναλωτής περιμένει κάποια δικαιώματα διευκολύνσεις ε, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ε, ο επιχειρηματίας, ο, ο τουρίστας, ο καταναλωτής, ε, ο συνταξιούχος, ο ασθενής, όλοι κάτι περιμένουν ε, και μιλάω δηλαδή για μια κοινωνία στην οποία όλοι οι πολίτες σε διάφορες ε, φάσεις της ζωής τους περιμένουν μια βελτίωση. Πρόκειται για τον κοινό μας βίο, τον κοινό ευρωπαϊκό μας βίο Υπάρχουν κανόνες που πλαισιώνουν τον βίο αυτό, ε, είναι κανόνες που μας ενώνουν σε έναν κοινό χώρο. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κάπως απογοητευμένη αίσθηση. Ε, ε, ο Μάριο Μόντι μίλησε για την κατάσταση του πολίτη καταναλωτή και τη σχέση του με την εσωτερική αγορά και πρόκειται για ένα ζήτημα που θα με απασχολήσει κατά τα ερχόμενα πέντε χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω την αύξηση του ΑΕΠ, ε, την, τον επιπλέον πλούτο χάρη στον κοινό αυτό χώρο οικονομικού βίου και του αριθμού τον αριθμό των θέσεων απασχόληση. Υπάρχει όμως ε, ένα χάσμα στις προσδοκίε, ε, μεταξύ δηλαδή χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και των 1.400 ε, οδηγιών που αφορούν την εσωτερική αγορά. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα στις 13 Ιανουαρίου και σας το λέω και σήμερα, η φιλοδοξία μου είναι να δώσω μια νέα όθηση σε αυτήν την ενιαία, στην, την εσωτερική αγορά. Και για να απαντήσω και σε μια ερώτηση του Προέδρου ε, Χάρμπορ, ε, η νέα αυτή όθηση είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής ε, της οικονομικής. Ναι, είναι η απάντησή μου, σαφέστατα. Η νέα αυτή όθηση είναι, έχει φανεί ήδη ως άξονας της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2020 θα είναι η προτεραιότητα σε όλες ε, τις ε, ε, πτυχές της στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, βέβαια στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με τους κοινωνικούς εταίρους, με τις περιφερειακές αρχές και με τους ίδιους τους πολίτες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις βασικούς τομείς, πριν ακούσω τις ερωτήσεις σας, για το νομοθετικό πρόγραμμα. Πρώτον, από τους κανόνες ε, στα δικαιώματα. Πρέπει να εφαρμοστεί η κοινοτική νομοθεσία. Υπάρχουν οι κανόνες, χρήσιμοι είναι, πρέπει όμως να εφαρμοστούν σωστά, πρέπει να γίνουν, να γίνουν κατανοητοί και να χρησιμοποιούνται σωστά. Κάθε εθνική ε, διοίκηση, περιφερειακή ή τοπική, έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει στην εφαρμογή Τη μία ή τη άλλη μεταξύ των 1.400 οδηγιών, μεταξύ των 1.400 κειμένων για, τις οποίες, ε, για τα οποία είμαι υπεύθυνο. Πρέπει λοιπόν για να εφαρμοστούν αυτά τα κείμενα να έχουμε περισσότερα μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλές προσφυγέ για παραβιάσεις, ε, όπως ε, για παράδειγμα ο κ. Μπουζόη για το Solvit ε, ε, συνέταξε μία έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερος διάλογος μεταξύ των ε, εθνικών και των περιφερειακών διοικήσεων. Πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την ευρωπαϊκή αριστεία στον τομέα αυτό, δηλαδή μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες για την οποία μιλήσαμε χθε, την οποία παρακολουθεί η κυρία Γκέπχαρτ και πολλοί από εσά εφαρμογή για, της για τα επαγγελματικά επιχειρηματικά ε, προσόντα, το σύστημα πληροφόρησης εσωτερική αγοράς, το IMI, να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιο είδους Facebook της εσωτερικής αγοράς, ε, ε, στο οποίο οποιαδήποτε, για όποια οδηγία και να μιλούμε, η εθνική ή η περιφερειακή διοίκηση μπορεί να συνεργάζεται με άλλες, ε, να ανταλλάσσει απόψεις για να μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα οικονομικών εταίρων ε, ή πολιτών. Βρίσκομαι λοιπόν στο ίδιο μήκο κείμενο ε, κύματο με τον Λουί Γκρέσ για μια πραγματιστική, για μια ρεαλιστική προσέγγιση την οποία χρειαζόμαστε. Όπως για παράδειγμα η ιδέα του εντοπισμού των, των των βασικών προγραμμάτων, των ε, βασικών 20 προγραμμάτων, του top 20 των προγραμμάτων, εν πάση περιπτώσει, που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών σε καθημερινή βάση. Ένα φόρουμ, ε, λοιπόν, ε, προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαμε να συναντιόμαστε, γιατί όχι εδώ στο Κοινοβούλιο, τακτικά, για να συζητούμε τα θέματα που αφορούν τους πολίτες στο, στο πλαίσιο δηλαδή την κοινωνία των πολιτών να έχουμε συγκεκριμένους στόχους, να τους αξιολογούμε, να, έχουμε, να κάνουμε μια συγκριτική αξιολόγηση ε, και να βλέπουμε και τις ε, βασικές ε, αδυναμίες που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά. Θα ήθελα επίσης να υπάρξει μια χάρτα εσωτερικής αγοράς για τους χρήστες, δηλαδή μια χάρτα δικαιωμάτων των χρηστών ε, η Κομισιόν βέβαια δεν μπορεί να είναι η μόνη που θα συντάξει ε, τη συγκεκριμένη ε, χάρτα. Πρέπει να είναι ένα τμήμα ολόκληρων, ένα τμήμα των συνεδριάσεων στο πλαίσιο αυτού του φόρουμ που σας ανέφερα. Ελπίζω τον Ιούνιο του 2011 στην αρχή της Πολωνικής Προεδρίας να γίνει κάτι τέτοιο. στον μεγάλο αυτό ευρωπαϊκό χώρο τον επιτρέπει κανείς στον πολίτη να διαμένει κάπου αλλού, να σπουδάζει κάπου αλλού, να εργάζεται κάπου αλλού, ε, αποτελεί μια επιταγή πολύ σημαντική. Οι γραπτές ερωτήσεις ε, που λαμβάνω εκ μέρου σας ε, δείχνουν ότι αυτή είναι μια βασική ανησυχία σας. Το θέμα της οδηγίας της αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων έχει ολοκληρωθεί σχεδόν σήμερα και γνωρίζω ότι δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση και την ισοδυναμία των επαγγελματικών προσόντων, για παράδειγμα γλωσσικέ απαιτήσει που υπάρχουν, ενδεχομένω καλέ ιδέε όπω ε, η, η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Χάρτα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Η κυρία Βερνιό θα με βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή και γι' αυτό ακριβώ οι υπηρεσίε μου έχουν δρομολογήσει παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγηση. Ερχόμαστε σε επαφή με διάφορου ε, ενδιαφερόμενους φορείς ε, καθ' όλη τη διάρκεια του 2010. Είναι πολύ σημαντικό να τροποποιήσουμε την συγκεκριμένη οδηγία και θα προτείνω στις αρχές του 2012 μια αναθεώρηση. Ένα ακόμη ζήτημα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενδιαφέρονται πάρα πολύ ε, είναι οι υπηρεσίες κοινή ωφελίας. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, υπηρεσίες, που πρέπει να παρέχονται, που είναι συχνά απομονωμένες, ε, δεν βλέπουν πολύ καλά σε τι τους εξυπηρετεί η Ευρώπη και συγκεκριμένα η εσωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε μια οδηγία πλαίσιο ευρωπαϊκή, όπως ε, κάποιοι από εσά ε, θα ήθελαν. Χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο, χρειάζεται τομεακή προσέγγιση. Πολύ ειλικρινά θα σας απαντήσω, δυόμιση χρόνια μετά την ε, ανάληψη καθηκόντων μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να προστατεύσουμε τις, τις δημόσιες υπηρεσίες, ε, τις υπηρεσίες κοινή ωφελία. Αυτό είναι απολύτω βέβαιο και τις πιο αδύναμες υπηρεσίες της κοινωνίας μας ε, πρέπει πάση θυσία να το κάνουμε αυτό. Στο, στο, στην περίπτωση, για παράδειγμα, της απελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών ε, θα συναντήσω αύριο τους ε, εταίρους ε, που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης, λοιπόν, των ταχυδρομικών υπηρεσιών πρέπει η αρχή της οικουμενικής υπηρεσίας που ορίζει ο κανονισμός να διατηρηθεί και να τύχει σεβασμού. Όπως και να έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, ε, η δική μου εντολή, δική μου, το δικό μου καθήκον είναι να έχουμε υπηρεσίες κοινή ωφελία ποιοτικέ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτές οι υπηρεσίες ε, είναι οι, αυτές που δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να ασκήσει τα βασικά του δικαιώματα. Οι πολίτες ε, για τους οποίους ε, μιλώ πάρα πολύ γιατί ακριβώς ε, αυτούς έχω συνεχώς στο μυαλό μου περιμένουν πολλά για να μπορούν να δουν τα δικαιώματά τους ε, να υπάρχουν στην καθημερινή τους ζωή, να μπορούν να τα ασκούν, ε, δυνατότητα πρόσβαση σε βασικές ε, υπηρεσίες, σε καλές τραπεζικές υπηρεσίες για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει την, τα δικαιώματά του ο πολίτης, ε, προβαίνει σε πώληση των ε, εμπορευμάτων του, για παράδειγμα, πρέπει να μπορεί να το κάνει με διαφανή και τίμιο τρόπο. Η εσωτερική αγορά είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικό, έτσι το βλέπω εγώ. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και να λάβουμε υπόψη και άλλα ε, στοιχεία. Για παράδειγμα, το φθινόπωρο, εγώ θα προτείνω στο Σώμα των Επιτρόπων διάλογο για τα παιχνίδια online θα το συζητήσω ε, όλος ιδιαίτερο το φθινόπωρο. Η συγητή σας με βοήθησε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για την ανάπτυξη της ε, ευρωπαϊκής δραστηριότητας ε, όσον αφορά τον ανταγωνισμό που είναι πάρα πολύ έντονος. Νομίζω υπάρχουν 15.000 ε, παράνομα sites αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας που ενθαρρύνουν την κατάσταση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι η καταπολέμηση ε, της ε, εξάρτησης, η προώθηση της κοινωνικοπολιτιστικής δραστηριότητας, η ενθάρρυνση των νέων είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Η οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντική επίση. Οι επενδύσει είναι ο μοχλό τη οικονομία και η εσωτερική αγορά πρέπει να ε, αναλάβει το ρόλο της και αναφέρομαι στις υπηρεσίες που είναι τα δύο τρίτα της ευρωπαϊκής οικονομίας ε, και σας το λέω όπω σας το είπα και χθε. Μία από τις προτεραιότητες μου είναι η εφαρμογή των, ε, ε για τις υπηρεσίες από 0,5 ως 1,5% επιπλέον θα ήταν το οικονομικό όφελος από την καλή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και θα επανέλθω στην Επιτροπή σας για να παρουσιάσω τα ε, αποτελέσματα αυτής της αμοιβαίας αξιολόγησης μεταξύ των κρατών μελών ε, και βάσει αυτών θα δούμε κατά πόσο πρέπει να επεκτείνουμε την ρητή η ε, στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 πρέπει να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση της ε, ε ευφυΐας και της καινοτομίας. Ε, για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η οι καινοτομίε και ε, όλες οι δημιουργικές πρωτοβουλίες πρέπει να αμείβονται ε, σωστά και δίκαια. Οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις ε, έχουν το δικαίωμα να περιμένουν νομοθετικό πλαίσιο πιο ευνοϊκό για αυτές. Δέκα φορές είναι πιο ακριβό, ακριβή μια έβριση τεχνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ΗΠΑ για για ποιο λόγο, αυτό για μένα είναι μια πολύ σημαντική, προ... το... μια πολύ σημαντική προτεραιότητα και είμαι σίγουρος και για την Ισπανική Προεδρία αυτή τη στιγμή, το ζήτημα της ευρωπαϊκής ε, ευρεσιτεχνίας. Πολλές φορές ε, το έχω συζητήσει και μαζί σας. Ε, σε ένα μήνα θα παρουσιάσω μία πρόταση για το γλωσσικό καθεστώς. Όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού, πρέπει να επιτρέψουμε και στο δημιουργό και στους χρήστες να ορίσουν οικονομικά μοντέλα βιώσιμα και στο διαδίκτυο, όσο υπάρχει νομικό περιεχόμενο, τόσο περισσότερο, περισσότερα είναι τα έσοδα αλλά παράλληλα πρέπει να καταπολεμήσουμε την πειρατεία και είναι γεγονός ότι η πειρατεία σήμερα αποδυναμώνει κάθε είδους ε, οικονομική αρχή, ε, όπως ε, για παράδειγμα μας είπαν οι Πολωνοί ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ σε μερικές υπηρεσίες Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το, το, το, το φθινόπωρο θα παρουσιάσω τις σχετικές προτάσεις. Πρέπει να δούμε επίσης την αναθεώρηση το 2011 της σχετικής οδηγίας ε, για τις υπηρεσίες ε, ε, που αφορούν τους δημιουργούς. Ο Ανδρέας Σφάμπ μου έδωσε την ιδέα μιας ευρωπαϊκής εκστρατείας για να εξηγήσουμε ακριβώς ε, πώς ε, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν κάθε όφελος να αγοράζουν νομίμως ε, για να προστατεύουν τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Βέβαια και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συμμετέχουν στη σχετική συζήτηση η εποπτεία επίσης ε, των αγορών λιανικής πώλησης ε, πρέπει να αξιολογηθεί ε, για παράδειγμα στον τομέα της διανομής. Πώς να εξηγήσουμε ότι τα υφάσματα κοστίζουν περισσότερο στην Ουγγαρία και, και, όχι στην, και, λιγότερο στην, στη Μεγάλη Βρετανία. Όταν ενδεχομένως υπάρχουν περισσότερα περιβαλλοντικά πρότυπα ε, που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ παραγωγών και μεγάλων αλυσίδων ε, διανομής. Στην άλλη πτυχή του χαρτοφυλακίου που με απασχολεί ε, μακρόν, γιατί ξέρετε ότι μας ενδιαφέρει μία σωστή χρηματοπιστωτική εποπτεία Υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά. Λίγες μέρες πριν ανέφερα στο Λονδίνο ότι θα πρέπει να χτίσουμε μία νέα δύναμη και ανταγωνιστικότητα. Όταν τα θεμέλια δεν είναι υγιή, αυτό θα έχει επιπτώσεις παντού. Και η χρηματοπιστωτική αυτή βιομηχανία ε, επιδεικνύει μεγάλη φαντασία, δηλαδή πολύ περισσότερη από ό,τι θα έπρεπε πολλές φορές ως προς τα προϊόντα που πολύ προς τον ε, καταναλωτή. Αυτή η βιομηχανία λοιπόν θα πρέπει να χτιστεί πάνω σε υγιή ε, θεμέλια. Οι G20 αποτελούν την οδική μας χάρτα μπορούμε να χτίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020. Μπορούμε να χτίσουμε την εσωτερική αγορά εκ νέου. Μπορούμε να άρουμε τα προσκόμματα ως προς την ψηφιακή οικονομία. Αλλά όλα αυτά δεν θα είχαν νόημα αν επέλθει μια νέα κρίση όχι μόνο επειδή ο φορολογούμενος πια δεν διαθέτει χρήματα και δεν, μπορεί να επιβαρυνθεί, δεν μπορούν να επιβαρυνθούν οι κρατικοί προϋπολογισμοί μια νέα κρίση, αλλά γιατί κανένας δεν μπορεί να υποστεί ένα νέο τέτοιο χρηματοπιστωτικό σοκ. Γι' αυτό χρειάζομαι τη βοήθειά σας γιατί εσείς είσαστε συνομοθέτες μέσα στα πλαίσια αυτού του εποπτικού έργου. Θα πρέπει να προωθήσουμε την πραγματική οικονομία και όχι την εικονική. Θα πρέπει να υπηρετούμε την πραγματική οικονομία. Αυτή την οικονομία θα πρέπει να υπηρετούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές σε πιο υγιή θεμέλια από αυτά που είδαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Θα ήθελα επίσης σε σχέση με την πραγματική ε, οικονομία να μιλήσω για το ρόλο των δημοσίων αρχών. Μιλήσαμε για την πρόθεση της καινοτομίας, της αηφόρου ανάπτυξης και της ε, καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα διασαφηνίσουμε με ένα συγκεκριμένο νομοθετικό έργο αυτούς τους στόχους για την, ε, για την ε, αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάθε μορφή εταιρικότητας και συνέργεια δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Ξέρω ότι η Επιτροπή το 2006 με την έκθεση Βάιλερ άνοιξε αυτό το δρόμο. Η τελική έκθεση δεν έχει εγκριθεί, αλλά πρόκειται για προστιθέμενη αξία η οποία προωθείται. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια καλή ρύθμιση και βεβαίως η Κομισιόν θα πρέπει να αποδείξει την προστιθέμενη αξία αυτής της ενδεχόμενης νομοθεσίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη την οικονομική ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων και νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει νομική ασφάλεια και διαφάνεια μέσα στα πλαίσια μιας ενδεχόμενης πρωτοβουλίας η οποία επακριβώς θα λάβει υπόψη την ανάλυση αντικτύπου που θα διενεργηθεί το 2010. Ως προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτή είναι μια άλλη προτεραιότητα, έχει μεγάλη σημασία το διασυνοριακό εμπόριο σε 23 κράτη-μέλη που αποτελεί κάτω από το 2% των λιανικών πωλήσεων. Η έκθεση Ετσεβαρία τόνισε τις ρίζες της κακοδαιμονίας και αυτό που έχει σημασία είναι και οι ηλεκτρονικές τιμολογήσεις μέσα στα πλαίσια του ΣΕΠΑ. Και αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε ε, ένα σωστό σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών online, έτσι ώστε να έχουμε μία ευφυή και αηφόρο ανάπτυξη. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι η διασυνδεσιμότητα ως προς τα ε, διάφορα δίκτυα και αυτό αφορά και τον τομέα του καμποτάζ ο οποίος θα μας απασχολήσει. Έχει μεγάλη σημασία να κινητοποιηθούμε συλλογικά ως Κομισιόν, 17 επίτροποι από τους 27 ασχολούνται με την καλή εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και θα προσπαθήσουμε να άρουμε κάθε πρόσκομα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε την, ε, τις διαστάσεις αυτές της εσωτερικής αγοράς. Επειδή είμαι ανοιχτός προς τα έξω, με ενδιαφέρει και η εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς ως προς τις δημόσιες προμήθειες, έσω και έξω. Αυτός είναι ο πυκνός οδικός χάρτης που έχουμε ενώπιον μας για να ξεπεράσουμε αυτή την κόποση την οποία ζούμε και να δώσουμε μία νέα όθηση, να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και της εσωτερικής αγοράς. Αναμένω με αδημονία την έκθεση του Μάριο Μόντι για να δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με το αρχικό μας ε, όραμα που εξεφράστη το 85 από τον Ζακ ε, Ντελόρ. Θα δω ποια θα είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης Μόντι και βεβαίως τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό μέσα στα πλαίσια μιας ανακοίνωσης. Θα ήθελα να γίνει ευρία διαβούλευση με όλους τους φορείς για να αναλάβουμε αυτή τη νέα συλλογική δέσμευση, αυτή τη ε, λευκή βίβλο. Ο Malcolm Harbour μίλησε για το Single Market Act, για την πράξη της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε το περιεχόμενο και μετά την ε, σωστή ε, επωνυμία. Αυτό το εγχείρημα ε, ξεπερνά το δικό μου χαρτοφυλάκιο υπό την στενή έννοια και γι' αυτό μου ζητήθηκε να προωθήσω αυτή την εργασία με όλους τους επιτρόπους που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία μέσα στα πλαίσια του Single Market Act διότι μιλάμε για μια νέα φιλοδοξία για την εσωτερική αγορά. Και βεβαίως θέλω να ακούσω και τη δική σας γνώμη, τη γνώμη της Επιτροπής σας εκ νέου. Σας ευχαριστώ πολύ. Well, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι απόλυτα σαφές το πώς ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της εργασίας της Κομισιόν για το 2010 θα εμπέσει στα δικά σας ε, καθήκοντα και κατανοείτε κι εσείς ότι παρόλο που η ε, γνωμοδότηση του καθηγητή Μόντι όντω μιλά για κούραση της ε, ε, εσωτερικής αγοράς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει καμία κούραση στην εδώ Επιτροπή τουλάχιστον, γιατί βλέπουμε πόσος μεγάλος είναι ο αριθμός των εκθέσεων. Η κυρία Ρούιλε, άλλοι συνάδελφοι έχουν υποβάλει γνωμοδοτήσεις για το κλειδιά, η κυρία Γκέφχαρτ για την μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες και πολλές άλλες που θα συνεχίσουμε να ε, επί των οποίων θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα και με, μεγάλη, με μεγάλο κέφι. Για του συναδέλφου που δεν ήταν εδώ στην αρχή, χαίρομαι που είμαστε πολλοί αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Να σα ε, θυμίσω ότι ε, σήμερα μιλούμε για το πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν για το 2010. Οπότε, αν μπορείτε, επικεντρώστε και τα ερωτήματά σα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στου συντονιστέ όλων των ομάδων να πάρουμε τρεις-τρεις τις ερωτήσεις αυτές και σας παρακαλώ να είσαστε και λίγο σύντομοι, συνεκτικοί για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια συζήτηση. Θα δούμε τώρα πώς θα πάμε από χρόνο. Σας παρακαλώ πάντως να είσαστε σύντομοι και να συγκεντρωθούμε στο συγκεκριμένο θέμα και όχι να μιλούμε γενικώ. Λοιπόν, η κυρία Σφάμπ, ο κύριος, η κυρία Γκέφχαρτ και μετά ο κύριος Μπουζόη. Κύριε Σφάμπ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά Επίτροπε, θα είμαι σύντομο ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να αναφέρουν τις παρατηρήσει τους. Σε πέντε βασικά σημεία θα επικεντρωθώ. Δικαίως είπατε, κύριε Επίτροπε, ότι ο πρώην ε, ε, Επίτροπος ε, Ανταγωνισμού Ομόντι μίλησε για κούραση της εσωτερική αγορά. Και βλέπουμε τώρα τι μπορεί να συμβεί με αυτή την κούραση που οδηγεί σε ανενεργία τους συμμετέχοντες. Βλέπουμε τι γίνεται σήμερα με την Ελλάδα. Τι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν τα κράτη-μέλη είχαν ε, εφαρμόσει από κοινού το πακέτο σταθερότητας, το σύμφωνο σταθερότητα. Τώρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο να μην πάνε καλά τα πράγματα. Ελπίζω να υπάρξει νέα όθηση για την εσωτερική αγορά, η οποία όχι μόνο βοηθά τις επιχειρήσεις, αλλά και τους πολίτες. Γι' αυτό εμείς ως ΕΛΚ θέλουμε να ε, θεωρούμε την, ε, να βλέπουμε την ε, εσωτερική αγορά από την πλευρά των πολιτών. Για παράδειγμα, στα πλαίσια τη ενιαία αγορά και τη πράξη για την ενιαία αγορά, που θα ψηφίσουμε αργότερα γιατί ένα κομμάτι το έχει συντάξει και ο κύριος Γκρέκ, έχουμε θέσει το θέμα των υπηρεσιών κοινού συμφέροντος. Και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι δεν χρειαζόμαστε οδηγία πλαίσιο, και η αιτιολόγηση αυτών των υπηρεσιών που ε, προσφέρει ο δημόσιος τομέας πάντα πρέπει να απευθύνεται στους πολίτες, να ασχολείται μόνο εάν, να υφίσταται εφόσον υπάρχει ανάγκη που προκύπτει από τους πολίτες. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε και νομικώς να τους εξασφαλίσουμε. Γι' αυτό χαίρομαι για αυτό που είπατε σχετικά. Να έχουμε δηλαδή μια τομεακή προσέγγιση και να βρούμε έτσι λύσει. Γιατί έτσι θα μπορέσουν να τι χρησιμοποιήσουν καλύτερα και οι πολίτε. Δεύτερον, θέσατε το θέμα του τι μπορούμε να κάνουμε στην εσωτερική αγορά σε ό,τι αφορά την απασχόληση, τι θέσει εργασία που εξασφαλίζονται μέσω τη εσωτερική αγορά, να δούμε ποιε είναι οι πρωτοβουλίε που υπάρχουν και μέσω του φόρουμ. Θα μπορούσαμε όντω να δούμε τι γίνεται και με τα παραποιημένα προϊόντα για τα οποία δυστυχώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να αντιμετωπίσουμε λοιπόν πιο ενεργά το θέμα αυτό και μέσω δημοσίων ε, εξαρτιών και ενημέρωση. Επίσης, είπατε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ε, ε, τομεακή προσέγγιση και για το νοχικό δίκαιο. Και γι' αυτό πρέπει ο δημόσιο τομέα, μιλήσατε κι εσεί και είπατε ότι όλοι και οι τοπικοί φορεί και οι περιφερειακέ αρχέ συμμετέχουν στην εσωτερική αγορά πάει με γνώμονα το καλό των πολιτών. Αυτό λοιπόν πρέπει να προωθηθεί και σε ό,τι αφορά τι ανταγωνιστικέ υπηρεσίε και αυτό πρέπει να γίνει και σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο να υπάρχουν, ε, να υπάρχουν διαγωνισμοί κλπ. Τέταρτον, συνέπειε τη τραπεζική κρίση στου καταναλωτέ στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό ε, να δούμε τι θα γίνει και με τη ρύθμιση των τραπεζικών αγορών πρέπει να θέσουμε κάποια σημεία τα οποία να είναι προ όφελο, να ρυθμίζουν τι τράπεζε και να είναι προ όφελο των καταναλωτών και των πολιτών. Γιατί πραγματικά και αυτοί πρέπει να εξασφαλίσουν ότι α, θα, οι επενδύσει του θα είναι εξασφαλισμένε. Θα σας, ε, μπορώ εγώ να σας εξασφαλίσω πάντως και να σας βεβαιώσω ότι θα έχετε το ΕΛΚ στο πλευρό σας, εάν όντως θέλετε να τα εφαρμόσετε όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστώ, η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπαρνιέ Χαίρομαι που το ξαναβλέπουμε σήμερα εδώ, γιατί τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσουμε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο συνέχεια μας θέτουν οι πολίτες. Τι μας δίνει η Ευρώπη. Αυτό μας θέτουν συνέχεια ως ερώτημα. Και πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια εσωτερική αγορά για τους πολίτες, μια, μόνη, μια ενιαία αγορά, εσωτερική αγορά, όπω και να την πείτε, πράξη για την ενιαία αγορά. Τέλο πάντων το σημαντικό είναι να μπορούν οι πολίτε να αναγνωρίσουν ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι για αυτού. Όχι για την οικονομία, όχι για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όχι για τι υπηρεσίε μόνο. Να είναι κάτι που να απευθύνεται σε αυτού για να μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια. Προ το παρόν αυτή την εντύπωση δεν την έχουν οι πολίτε. και πρέπει να το, να το διορθώσουμε αυτό. Δέχομαι και η ομάδα μου επίσης ότι ως πρώτη προτεραιότητα θέτεται τα προβλήματα τη της οικονομικής κρίσης και ότι θέλετε να δεσμευτείτε, να εμπλακείτε όσο το δυνατόν περισσότερο στον τομέα αυτό, σε ό,τι αφορά βέβαια τι συνέπειε που έχει η οικονομική κρίση στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι ένα κομμάτι του του προγράμματο εργασία τη Κομισιόν. Εμεί ευχαρίστω να σα βοηθήσουμε στην προσπάθειά σα στου τομεί αυτού που είναι σημαντικοί να συνεχίσετε δηλαδή έτσι όπως ε, έχετε ξεκινήσει. Και βεβαίως ε, εδώ πρέπει να αναφέρουμε, αυτό που είπατε και εσείς βέβαια Επίτροπε, το πρωτόκολλο για την ε, συνθήκη της Λισαβόνας που αποτελεί και μια έτσι, οδηγία για την πολιτική της Ευρώπης, για τις υπηρεσίε κοινή ωφέλεια. Υπάρχει πολλή φόβο στου πολίτε, υπάρχει ανησυχία, ανασφάλεια και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Επίση, κάτι άλλο που είπατε και που είναι πολύ σημαντικό είναι όντω η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Γιατί έτσι μιλούμε για πρόσβαση σε, άλλες, σε αγορές άλλων χωρών. Και ε, εν μέρη υπάρχει καλή νομοθεσία, αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας χωλαίνει. Εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα. Και ακόμη και χτες το είδαμε στην ε, ακρόαση για την ε, οδηγία και τις υπηρεσίες. κάποιοι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια το ανέφεραν αυτό. Πρέπει λοιπόν πραγματικά κάτι να κάνουμε. Τρίτο και τελευταίο. Υπάρχουν και άλλα βέβαια που θα ήθελα να πω, αλλά θα επικεντρωθώ σε αυτά. Τα τυχερά παιχνίδια. Το είπατε κι εσείς, η κυρία Σόλτε Μόζε έχει κάνει πάρα πολύ καλή έκθεση για το θέμα αυτό και επί τη βάση αυτή πρέπει να κάνουμε κι εμεί κάποιε σκέψει για το πώ θα προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. Γιατί χρειαζόμαστε, ε, πρέπει να ε, προστατεύσουμε τους πολίτες έναντι της οργανωμένης εγκληματικότητας. Ε, εθνικός πώς μπορεί να κάνει καλυνής πολλά πράγματα και καλά. Αλλά όταν μιλούμε για τυχερά παιχνίδια στο ίντερνετ ας πούμε, σε μεγάλα δίκτυα, τότε εκεί χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή απάντηση, ευρωπαϊκή δράση. Και πιστεύω ότι ε, πρέπει να κινητοποιηθούμε προς αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι επίγον να κάνουμε κάτι. Γιατί εδώ μιλούμε για τους πολίτες μας, οι οποίοι διακινδυνεύουν παίζοντας σε τέτοια παιχνίδια. Και τώρα αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ρυθμιστεί αυτό. Πραγματικά νομίζω λοιπόν ότι για να μην σας πω για παγκόσμια λύση, τουλάχιστον ευρωπαϊκή λύση πρέπει να βρούμε σε αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Γκέπχαρτ. Ο κύριος Μπουζόη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Euh, en concernant le programme de travail que je considère. Εάν λάβουμε υπόψη το πρόγραμμα εργασιών, quelques initiatives liées au commerce électronique, e-commerce. Euh, papier vert euh, sur e-procurement. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες και το e-invoicing, δηλαδή τις ηλεκτρονικές τιμολογήσεις. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να δούμε τις, ε, τα δεδομένα της ενιαίας αγοράς έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην παγκόσμια αγορά. Αλλά όπως είπατε δεν είμαστε τόσο αποδοτικοί σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θεωρείτε ότι αυτό θα είχε μεγάλη επίπτωση στο εγγύς μέλλον. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος της εργασίας σας, το 10-11, σχετίζεται με αυτές, όχι μόνο με αυτές τις ε, καλές πρωτοβουλίες, αλλά και με την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Ήδη έχετε, νομίζω, ε, επισκεφθεί ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θεωρείτε ότι μιλάμε για πραγματική εφαρμογή της ε, νομοθεσίας και το πρόβλημα έγκυται στην, ε, στο γεγονός ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από ορισμένες χώρες ή θεωρείτε ότι έχουμε να κάνουμε με τεχνικές πτυχές εφαρμογής της νομοθεσίας. Ευχαριστούμε πολύ και υποστηρίζουμε την, το φιλόδοξό σας πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. Νομίζω ότι καταρχήν έχει σημασία να υπάρχει μια πραγματική ε, αμφίδρομη ακρόαση και θα προσπαθήσουμε να ε, προσδώσουμε σώμα σε αυτό το οικοδόμημα ε, βάζοντας ο καθένας ένα λιθαράκι κάθε φορά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι για την εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι υπάρχει Ευρώπη έναντι των πολιτών. Είναι μια διαρκής διαδικασία. Αυτό που έχει σημασία είναι δηλαδή να λάβουμε υπόψη ότι οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ε, θέλησαν να προσδώσουν οντότητα σε αυτή την πολιτική βούληση. Αυτό αφορά και την πεμπτουσία της ενίας αγοράς. Είναι η υλοποίηση των οικονομιών μας αλλά η διάρκεια αυτού του προγράμματος εδώ και 50 χρόνια πρέπει να μετουσιωθεί σε κάτι άλλο και γι' αυτό θα πρέπει να αποδείξουμε τις δυνάμεις μας. Θα ήθελα να πω στον Ανδρέα Σβάμπ ότι με τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και με τις περιφερειακές και τοπικές θα ήθελα να προωθήσω αυτό τον διάλογο και ιδιαίτερα με την κοινωνία των πολιτών και τις περιφερειακές κυβερνήσεις. Κύριε Σβάμπ, αυτό είναι ένα μείζον εγχείρημα. Και φυσικά μιλήσαμε για κόποση της Ευρώπης, αλλά μία από τις ανησυχίες των πολιτών αφορούν τις επιχειρήσεις γενικού ενδιαφέροντος. γιατί μιλάμε για 25% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30% απασχόλησης και υπάρχουν 500.000 φορείς που εμπλέκονται σε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Γι' αυτό ακριβώς ε, το θέμα αυτό σχετίζεται με την πεμπτουσία της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. Θα ήθελα με μεγάλη διάβγεια να δούμε αυτό το ζήτημα για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο. Θα υπάρχει μία μόνο διαπλαίσιο, όπως επιθυμούν οι σοσιαλιστές. Θα έχουμε τομεακές νομοθεσίες όπως θέλουν μερικοί, αλλά όχι παντού βεβαίως. Για άλλη μια μονο πλαισιο οπως επιθυμουν οι σοσιαλιστες θα πρέπει να εργαστούμε για να προστατεύσουμε τον πολίτη χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις, αντικειμενικά. Και αφού ακούσω τους πάντες, τότε θα διατυπώσω την τελική μου γνώμη. Υποστηρίζω πολλές πρωτοβουλίες που γνωρίζει και ο κύριος Σβάμπ υπέρ των καταναλωτών και θα προσπαθήσω να ε, ενσωματώσω στο πρόγραμμά σας και ε, και καθαρά οικονομικές συνιστώσεις. Διότι αυτή, μάλλον η μεγάλη ανησυχία των πολιτών σχετίζεται με την απασχόληση. Κυρία Γκέπχαρτ, υπάρχει απόσταση μεταξύ πολιτών και αγοράς. Γιατί οι πολίτες θεωρούν ότι η αγορά υπηρετεί τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – εγώ θέλω να δράσω υπέρ των ΜΜΕ και των καταναλατών και θα αναλάβουμε μια πράσινη πρωτοβουλία και για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα χρηματιστήριο των ΜΜΕ και περιφερειακά χρηματιστήρια τα οποία να, να προσανατολίζονται στην προσπελασιμότητα των ΜΜΕ προς αυτά προς αυτά τα περιφερειακά χρηματιστήρια, διότι αποτελούν το 80% της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ενιαίας αγοράς. Σας είπα πώς βλέπω το θέμα των δημοσίων αγορών και των δημοσίων προμηθειών. Εργαζόμαστε για την πράσινη αυτή βίβλο, για την αναγνώριση πτυχίων και διπλωμάτων. Είμαι πεπισμένος όμως ότι θα πρέπει να δράσουμε άμεσα, διότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο να απελευθερώσουμε τα τυχερά παιχνίδια και να τα στυλιτεύουμε. Αυτό το λέω ενώπιον του Κοινοβουλίου και το έχω πει κατά την ακρόασή μου. Δεν θα, ήθελα να απελευθερώσω τα πάντα και να στυλιτεύω εκείνους που δεν απελευθερώνουν την αγορά. Και αυτό αφορά και τα τυχερά παιχνίδια online, διότι υπάρχει και πρόβλημα εθισμού. Ε, εργάζομαι με την κυρία Κρές για ένα κοινό πρόγραμμα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Τώρα, κατά πόσο θα επέλθει η πρόοδος για το ηλεκτρονικό εμπόριο, Μα μιλάμε από έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Μιλήσαμε για ένα 2% του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ε, πιο κάτω δεν γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να επιτελεστεί πρόοδος στην εσωτερική αγορά και η κοινή ηλεκτρονική αγορά είναι ε, το μεγάλο αυτό οικοδόμημα το οποίο θα προωθήσουμε. Συνεργάζομαι με την Επίτροπο, την κυρία Κρές, και θα σας πούμε σε τι συμπεράσματα θα φτάσουμε. Κύριε Μπουζόη, δεν μπορώ να σας ε, δώσω σαφή απάντηση. Χτες μιλήσαμε για την οδηγία περί μαζί σας και για την μεταφορά της οδηγίας, η οποία δεν είναι παντού η ίδια. Άλλο μεταφορά, άλλο θέση σε ισχύ βεβαίως. Και αυτό αφορά και άλλες οδηγίες. Σε πολλές χώρες που δεν υπάρχει ένα τόσο συγκεντρωτικό σύστημα, τα πράγματα ίσως είναι πιο εύκολα. Γι' αυτό στις 3 Ιουνίου στην Στοκχόλμη θα αρχίσω ένα γύρο των πρωτεύουσών έτσι ώστε οι αρμόδιοι υπουργοί να με διαφωτίσουν και να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και οι αξιωματούχοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της οδηγίας όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, γιατί οι δημόσιες προμήθειες είναι το 17% του ΑΕΠ και πολλές φορές προωθούνται από τις περιφερειακές αρχές. Θα μιλήσω με τους υπευθύνους πριν περάσουμε σε ένα καθαρά κυρωτικό σύστημα. Θα δω λοιπόν πού υπάρχουν δυσκολίες και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να ε, μάθουμε από εσά τι θα γίνει, γιατί ανησυχούμε και εμείς. Λοιπόν, συνάδελφοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε τρεις ε, συντονιστές ακόμα. Θέλω να ακούσω και από τις ε, πολιτικές ομάδες, δηλαδή από όλους τους συντονιστές. Μακλάκεν, και ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι ο τρίτος. Μετά υπάρχουν τες, δέκα ομιλητές. Αφού, μας, ε, αφού απαντήσουν οι συντολιστές θα λάβετε το λόγο ένα λεπτό. Μία ερώτηση προς τον κύριο Μπαρνιέ ή κάτι που ε, υπολείπεται για ένα λεπτό, αυστηρά. Mr. Manders, Mr. Mrs. Mr. Abad, Mr. Θα έχετε λοιπόν από ένα λεπτό να θέσετε τα θέματά σας στον Επίτροπο, ώστε να έχει και ο Επίτροπος ε, χρόνο να σας απαντήσει, έτσι. Οπότε, να σας θυμίσω, συνάδελφοι, ότι στις 10 και 4 έχουμε ψηφοφορία, η οποία θα μεταδοθεί και στην τηλεόραση βλέπω και τις κάμερες εδώ. Σας παρακαλώ, ε, ελπίζω να έχετε φέρει τις ε, κάρτες ψηφοφορίας σας. Αν δεν τις έχετε, στείλτε κάποιον να τις πάρει. Η κυρία Ρουιλέ πρώτα για τον επόμενο γύρο των ερωτημάτων. Παρακαλώ. Κύριε Μπαρνιέ, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τι παρατηρήσει σα και χαίρομαι που είπατε ότι πρέπει η εσωτερική αγορά να έχει στόχο και σκοπό και δεν υπάρχει έτσι αυτόνομα και μόνο για να υπάρχει. Και θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία. Φυσικά θέλουμε να υπάρχουν όλα αυτά, θέλουμε να υπάρχει εκπαίδευση, αλλά υπάρχει και ένα θέμα καινού που είπατε μεταξύ τη εσωτερική αγορά και, και των πολιτών. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με, με το θέμα τη νομοθεσία. Στον τομέα αυτό και κυρίως στους τομείς τους οποίους, με τους οποίους ασχολούμαι εγώ έχουμε θέματα παραβίασης δικαίου, έχουμε πρωτογενές δίκαιο από την Κομισιόν το οποίο την χάνει πολλών ερμηνεών και όταν βλέπω εγώ το πρόγραμμα της Κομισιόν βλέπω ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ε, μη νομοθετικών πρωτοβουλειών soft law πρωτοβουλίε. Ε, αυτό εγώ το βρίσκω προβληματικό. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να σας, να σας πω και νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ασχολείται λιγότερο με το soft law και να ξεκινήσει ε, περισσότερες ε, ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες και να τις κοινοποιεί πολύ περισσότερο. Και επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερο εντο, συντονισμός εντός της Κομισιόν. Αυτό μου το βλέπω συνέχεια και ειδικά όταν έκανα την γνωμοδότηση για τις δημόσιες προμήθειες πάλι η Κομισιόν πέρασε στο soft law είτε γιατί δεν μπορούσε να συντονίσει, είτε μπορούσε να συντονίσει πολύ λίγο. Δηλαδή η μία υπηρεσία δεν ξέρει τι ερμηνεύει η άλλη υπηρεσία και πώ το ερμηνεύει. Νομίζω ότι αυτό είναι προβληματικό γιατί μετά δεν ξέρουν και οι υπόλοιπε, οι τοπικέ κοινωνίε, οι περιφερειακέ αρχέ δεν ξέρουν τι να περιμένουν. Οπότε πώ θα συντονιστούν αυτέ όταν δεν μπορείτε να συντονίσετε εσεί. Το θέμα του ενοχικού δικαίου έχει ε, είναι πολύ σημαντικό. Εμεί ω Κοινοβούλιο έχουμε λίγε γνώσει για το τι γίνεται μέσα σε αυτές τις εσωτερικέ επιτροπές και ξέρετε ότι είμαστε συνέχεια σε διαπραγματεύσει με την ε, Κομισιόν για τι επιτροπέ αυτέ. Πρέπει να μα δώσετε περισσότερε πληροφορίε. και θέλουμε πληροφορίε αυτέ που λαμβάνει και το, ε, και το Συμβούλιο. Θέλουμε να είμαστε επίση όρει. Επίση, μία παρατήρηση να κάνω για τι παρατηρήσεις που κάνατε για τις παραχωρήσει για τις υπηρεσίε. Πρέπει να μην χάσουμε από το στόχο μας τις κοινότητε. Πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση, ευρεία διαβούλευση και να αποφύγουμε να γίνει κατακαιρματισμό του δικαίου. Εγώ είμαι τη άποψη πριν φτάσουμε στο θέμα του ενοχικού δικαίου και προτείνεται νέα νομοθεσία ή νέο soft law, καταρχήν κάντε μία καταγραφή των πραγμάτων. Γιατί οι παρεξηγήσει που υπάρχουν στι κοινότητε και στο τοπικό επίπεδο πραγματικά οδηγούν σε τεράστια αδιέξοδα. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα, δεν μπορούμε να το ξεχνούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην πρώτη ακρόαση, Επίτροπε, με την Επιτροπή μας, είπατε ότι δεν θέλετε να επισκεφτείτε μόνο τις ε, πόλεις των κρατών μελών, αλλά και τις περιφέρειες. Χαίρομαι που θα το κάνετε. Ελπίζω να έρθετε και στη δική μου την περιφέρεια, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να αναφερθώ σε μια πρωτοβουλία που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε όλη την επικράτεια της χώρας και θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πώς θέλουμε εμείς να προχωρήσει όλο αυτό, ειδικά εισάγοντα μια νέα κάρτα εργασίας ευρωπαϊκή. Ελπίζω αυτό να γίνει άμεσα. Ευχαριστώ. Και τελευταίος, ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Κύριε Επίτροπε, σας άκουσα με πολύ προσοχή να υποστηρίζετε τη διατήρηση της ε, την ανάγκη για διατήρηση των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και την ανάγκη να τις ενισχύσουμε. Ωστόσο έχω μια ανησυχία μήπως η Επιτροπή προτίθεται να αλλάξει το χαρακτήρα και τη φύση των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, μειώνοντας ταυτόχρονα και το ρόλο του κράτους σε αυτές τις υπηρεσίες. Και το λέω αυτό κύριε Επίτροπε γιατί στην οδηγία για τις υπηρεσίες η έγκριση έγινε με τη σαφή εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής τη οδηγίας αυτή, των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή όμως έχει στα σχέδια της την ανάληψη μη νομοθετικών πρωτοβουλειών για την αναθεώρηση του πλαισίου των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Δεν είμαι σίγουρος πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέξει να ρυθμίσει τις όποιε εξαιρέσει από την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η ερώτηση μου είναι μήπως με ξεχωριστές οδηγίες που όμως θα αποτελούν παραρτήματα της συγκεκριμένης οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ο Επίτροπος να απαντήσει στις τρεις αυτές παρεμβάσεις και μετά θα έχουμε τις παρεμβάσεις ενός λεπτού από τους υπολείπους. Euh, Κυρία Ρούλε, σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες ε, διάβασα με μεγάλη προσοχή την έκθεσή σας και αναφέρομαι σε αυτή. Πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα η συνοχή είναι ύψης της σημασίας και αυτό αφορά την ε, Επιτροπή στο συλλογικό της έργο. Ήμουν επίτροπος υπεύθυνο για την περιφερειακή πολιτική στο παρελθόν υπεύθυνο για τον δεύτερο προϋπολογισμό των ε, ευρωπαϊκών κοινοτήτων της τάξης των 300 δις. Είχαν διαχειριστώ ένα προϋπολογισμό της τάξης των 300 δις. Με ενδιέφερε λοιπόν ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο πρόεδρος Ζακ Ντελόρ όταν ασχολήθηκε με την ενιαία πράξη ασχολήθηκε και με την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική για να μην υπάρχει περιφερειακός εδαφικός κατακαιρματισμός. Ζήτησα λοιπόν μαζί με τον κύριο Χαν στην γενική μας διεύθυνση να δούμε πώς οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν να εμπλακούν στην εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες ιδιαίτερα όταν υπήρχε κακοδιαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων ή η ε, ιδιαίτερη ε, περιπλοκότητα των κανόνων της εφαρμογής. Πρόκειται για, ε, πρόκειται για εσωτερική εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα τη συνεχίσουμε με τους νέους επιτρόπους. Θέλουμε να κάνουμε μία συνολική αποτίμηση της πλαισίωσης των δημοσίων προμηθειών μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2011 και το θέμα του soft law, της ήπιας νομοθεσίας, θα έχει μεγάλη σημασία έτσι ώστε να έχουμε ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να διευθετήσουμε αυτή την πλαισίωση των δημοσίων προμηθειών μέσα στα πλαίσια μιας ε, καινοτομίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, έχω αναλάβει πρωτοβουλίες ε, σε αυτό τον ε, τομέα. Κυρία Μακλάκιν, οπωσδήποτε θα παρέμβω σε περιφερειακό επίπεδο ε, δεν ξέρω πότε θα έρθω σε εσά, αλλά οπωσδήποτε θα μεταβώ στην πρωτεύουσά σας και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι θα γίνει επιτόπου σε κάθε περιφέρεια και όχι μόνο πρωτεύουσα. Ως προς τα επαγγελματικά προσόντα, κύριε Μακάρτιν, τώρα προβαίνουμε σε μία ε, αποτίμηση, αξιολόγηση της οδηγίας ε, για να δούμε και το γλωσσικό και το αργότερο το 2012 θα έχουμε μια τελική ε, έκθεση. Προσπαθώ όμως να κερδίσουμε χρόνο, να γίνει αυτό νωρίτερα ή δυνατόν. Σας είπα, ε, σκεφτόμαστε την κυρία Βερνιό και άλλους, ότι έχει σημασία να υπάρχει ε, μία επαγγελματική ε, κάρτα τουλάχιστον ε, για μερικά, αν όχι όλα τα επαγγέλματα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας είπα ότι θέλω να υπερασπιστώ αυτό το τομέα, πάση θυσία, και με ενδιαφέρει να δω ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση, δηλαδή τομεακή, αυστηρά τομεακή με μία οδηγία πλαίσιο ή με ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα στηριχτεί σε πολλά τομεακά κείμενα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το, το πρόβλημα στην φύση του πριν αποφασίσω για την προσέγγιση και όπως γνωρίζετε θα πρέπει να παγιοποιήσουμε και αυτή την έννοια των ε, δημοσίων ε, προμηθειών και στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ε, εισακούνται όχι μόνο οι Ευρωπαίοι βουλευτές, αλλά και οι Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις επί του θέματος. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο γιατί απαντήσατε πλήρως σε όλα τα σημεία των πολιτικών ομάδων. Τώρα θα αρχίσουμε με τις παρεμβάσεις ενός λεπτού. Ο κύριος Ζουβέ έχει ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σαφήνα τη παρουσίασής σας ε, και της γενικής θεώρησης της ε, εσωτερικής αγοράς που έχετε. Μιλήσατε για την οικονομική κρίση λέγοντας ότι αν ένα κράτος μέλος ε, έχει έλλειμμα ενδεχομένως μπορεί διακόπτη ο πρόεδρος. Παρακαλώ ή ησυχία κάντε ή αποχωρήστε γιατί κάνετε πολύ θόρυβο. Αν χρειάζεται να κάνετε διαπραγματεύσεις, όχι κάτι διάρκεια τη συνεδρίαση. Κύριε Ζουβέν, επιπλέον 30 δευτερόλεπτα έχετε για να συνεχίσετε. Ευχαριστώ. Δηλαδή 30 λεπτά παραπάνω μου δίνετε. ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι η οικονομική κρίση και η ζωτικότητα της εσωτερικής αγοράς συνδέονται και η επικαιρότητα μας το αν ε, ένα κράτος μέλος έχει αδυναμία πληρωμών ε, ολόκληρο το σύστημα θα ε, είναι ευαίσθητο, θα είναι βάλωτο. Αναφέρετε σε, αναφέρεστε σε δύο πράγματα. Αναφέρεστε στη σημασία της στρατηγικής αλλά και στη, στο γεγονός ότι η στρατηγική πρέπει να γίνει κατανοητή και σεβαστή από όλα τα κράτη-μέλη. Πιστεύετε ότι αυτή, αυτό ισχύει σήμερα. Είναι όλοι οι εταίροι επαρκώς ε, εμπλεγμένοι για να αντιμετωπίσουν μια κρίση όχι μόνο ελληνική αλλά ευρωπαϊκή. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζουβά. Ο κύριος Μάντος. Και μετά ο κύριος Γκρέκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρουσίασή σα. Για να βελτιώσουμε τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά, νομίζω ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε μόνο σε κανονισμού και όχι τόσο σε οδηγίες, γιατί αυτό είναι συνήθω το πρόβλημα, ότι ε, είναι διαφορετικό το επίπεδο σε κάθε κράτο μέλο, οπότε είναι κακή η λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Έχουμε πολλέ φορέ συζητήσει μαζί ε, το, το, το θέμα τη ευρεσιτεχνία. Ελπίζω να λύσετε το πρόβλημα το γλωσσικό ε, και μάλιστα στο πλαίσιο ενός κανονισμού και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και ένα πρόβλημα θα έχουμε και ένα ζήτημα επίλυσης ε, ε, διαφορών που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες έχω συγκεκριμένο ερώτημα. Έχω λάβει πάρα πολλά παράπονα επιχειρηματιών ε, και ε, καταστηματαρχών ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματά τους ε, σε μεθοριακές περιοχές τις Κυριακές, αλλά σε άλλες χώρες μπορούν να το κάνουν και αυτό το θεωρούν στρέβλωση της ελεύθερης κυκλοφορίας, της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα γιατί υπάρχει ασάφεια. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Μάντες, ο κύριος Γκρέκ και μετά ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας ε, και η κυρία ε, Βερνιό. Κύριε Γκρέκ. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι πρέπει να κάνουμε τη μετάβαση από τους κανόνες στα δικαιώματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ πιστικό ε, σλόγγαν, ε, ειδικότερα όταν θέλουμε να ολοκληρώσουμε, να βελτιώσουμε τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Ε, οι πολίτε δεν γνωρίζουν καλά πώ δουλεύει η εσωτερική αγορά, ούτε τα δικαιώματα, ούτε τα ωφέλη. Πώ θα μπορέσουμε να μεταφράσουμε το σλόγγαν αυτό που αναφέρατε σε μια συνεκτική στρατηγική μέχρι το 2012. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν και πάρα πολύ σύντομο, λέει ο πρόεδρο η κυρία Βερνιό, η δεύτερη αντιπρόεδρο, ε, και μετά ο κύριο Σαμπάρτο. Κυρία Βερνιό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα κόψω πολλά από αυτά που ήθελα να πω. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο γιατί έχει μία φιλοδοξία, αλλά έχει μία φιλοδοξία που εξυπηρετεί ένα όραμα. Πολλοί πολιτικοί έχουν φιλοδοξίες, αλλά όχι όραμα, οπότε θα συνεργαστούμε θα προσπαθήσω να, να επισημάνω τρία ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά και για μένα και για τους πολίτες. Ε, τονίσατε τη σημασία της χάρτας της Ευρωπαϊκής ε, για τα επαγγελματικά προσόντα. Είναι κατεπήγον αυτό το ζήτημα γιατί μια καλή λειτουργία της οδηγίας για τις υπηρεσίες έχει σχέση και με αυτό. Μιλήσατε επίσης για το θέμα της, ε, της, των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών κοινή ωφελίας. Μιλήσατε επίσης για για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο σεβασμό τη Οικουμενική υπηρεσία σε όλε τι δημόσιε υπηρεσίε, προστατεύοντα, γιατί μιλήσατε για προστασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι σπάνιο ο Επίτροπο Εσωτερική Αγορά να χρησιμοποιεί τον όρο προστασία. Αν οι πολίτες αισθάνονται προστατευμένοι στη δουλειά τους και στη ζωή τους, θα είναι πολύ πιο ικανοί στο πλαίσιο της εργασίας τους να καινοτομήσουν και να αναλάβουν ευθύνες. Ενδεχομένω, η οικονομία και η ανταγωνιστικότητα δεν θα είναι ταμπού για τα εκατομμύρια εργαζομένων ε, και έχουμε περάσει δύσκολε στιγμές, ειδικότερα στην ε, Γαλλία και στην Ολλανδία ε, το 2005. Και τελευταία μου παρατήρηση για τι τραπεζικέ υπηρεσίε, Μιλήσατε για διαφάνεια και για ενίσχυση στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικότερα για τα περιφερειακά χρηματιστήρια και αυτό είναι σημαντικό. Ε, θα θέλατε να μου πείτε τι προθεσμίες έχετε για, τα, για τις προτάσεις σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ο ρόλος των τοπικών ε, και περιφερειακών αρχών ε, και αυτός είναι πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ. μισή λεπτό για τρεις ερωτήσεις, κυρία Αντιπρόεδρε. Μπράβο σας. Ο κύριος και μετά ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Πίτροπε για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Μία ακόμη φορά, δύο ζητήματα. Μιλήσαμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες κοινή ωφελίας, είμαι ησυχητής για το θέμα αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερως που δίνεται μια πολιτική διάσταση στο ζήτημα αυτό, υπενθυμίζοντας απαιτήσει προστασία συνοχής και αλληλεγγύης, όπως επίσης το ρόλο κοινωνικού, ε, το κοινωνικό ρόλο που μπορεί να έχουν ε, τέτοιου είδους υπηρεσίες σε περιόδους κρίσεως, ε, ο πολιτισμό είναι πιο σημαντικό από την ιδεολογία και θέλω να μου πείτε το, σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται ε, η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν τα ζητήματα της επικουρικότητα είναι επίση πολύ σημαντικά και να μου πείτε και μερικά πράγματα για την ε, ε, ανακοίνωση της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει για αυτό το θέμα. Θα θέλω να μου πείτε επίσης ε, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες σας για να υπάρχει μια βιομηχανική πολιτική ε, ψηφιακή όπως ε, στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φάντερκαμπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο και για το πρόγραμμα που μας παρουσίασε, αλλά και για τις φιλοδοξίε του. Νομίζω ότι έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση από, τις φιλοδοξίες και ε, νομίζω ότι είστε ο σωστό άνθρωπος στη σωστή θέση, κύριε Μπαρνιέ. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, ε, την οδηγία για τις υπηρεσίες, ε, η πρώτη αναθεώρηση προβλέπεται για το Δεκέμβριο του 2010. Κάποιες χώρες όμως ε, δεν έχουν καν μεταφέρει την οδηγία αυτή στο εσωτερικό τους δίκαιο ακόμη. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτή την προθεσμία. Δεύτερον, η οδηγία για, το, για τις υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Ακούω πάρα πολλά παράπονα στη χώρα μου, στις κάτω χώρες, ότι δεν ε, έχουν ε, κάνει τα απαραίτητα ε, ορισμένες χώρες στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής ευρωπαϊκής της οδηγίας αυτής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επιτροπό. Πολύ ενδιαφέρονται αυτά που είπατε για την προστασία των καταναλωτών και τα οικονομικά προϊόντα. Φυσικά πρέπει να έχουμε άποψη ως προς αυτό, αλλά το, αυτό που είπατε για τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε πού ακριβώς θα μπει. Για μας τουλάχιστον είναι σημαντικό. Επίσης, όταν θα έρθετε να επισκεφτείτε τις περιφέρειες του, του Ηνωμένου Βασιλείου, ελάτε και προς τη Σκωτία. Έχουμε μεγάλο τομέα υπηρεσιών. Τώρα, για την εσωτερική αγορά, Ε, υπήρξε πρόβλημα ε, πολύ σημαντικό σαν αυτό με το, με το ηφαίστειο. Ε, τώρα με την Ισλανδία μπορεί το δεύτερο ηφαίστειο να είναι πιο καταστροφικό από το πρώτο που εξεράγει την προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τάιλερ. Η κυρία Ράπτη και μετά η κυρία Τούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ το περιεχόμενο και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάσατε το σχέδιό σας δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης όμως εκτός από τη θεωρία και τα πάρα πολύ ωραία λόγια υπάρχει και η πραγματικότητα και η πραγματικότητα λέει ότι για να χτίσουμε το 2020 όπως είπατε πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό το 2010, το 2011, το 2012, το 2013 και το 2010 η Ευρώπη δέχεται μία πίεση. Βιώνουμε μία οικονομική κρίση. Μιλάω για την ελληνική κρίση που έχει ευρωπαϊκή διάσταση και αυτό το βλέπουμε γιατί οι κερδοσκόποι εκτός από την Ελλάδα βάζουν τώρα στο στόχο και άλλες χώρες. Θυμίζω την επίθεση που, δέχτε, που δέχεται πλέον η Πορτογαλία από τους κερδοσκόπους. Πόσο λαμβάνετε υπόψη στους σχεδιασμούς σας αυτή την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και δεύτερον πώς προτίθεστε να προστατεύσετε τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ένα τέτοιο οικονομικό πλαίσιο που δημιουργείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ραπτή. Η κυρία Τούν και ο καθηγητής Κορέα Δεκαμπός μετά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν, Επιτροπέ, να σας ευχαριστήσω για την πολύ εντατική συνεργασία μας. Χαίρομαι να ακούω όλες αυτές τις προοπτικές που έχετε θέσει. Μιλήσατε για την καλή ε, συνεργασία που έχετε με άλλους ε, επιτρόπους, με άλλες υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφέρατε και ανοιχτά τα κράτη-μέλη. Ε, δίνετε λοιπόν μεγάλη προσοχή στα νέα κράτη-μέλη. Μερικές φορές δεν συμβαίνει αυτό όταν έρχονται να μας μιλήσουν κάποιοι άλλοι επίτροποι. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μιλήσατε για ένα ποσοστό 2% και η πειρατεία χρειάζεται μια μακρόπνοη ε, στρατηγική για την αντιμετώπιση της. Πρέπει φυσικά να βοηθήσουμε αυτούς που ε, μπορούν ή θέλουν να ε, αγοράσουν ηλεκτρονικά. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην στραγγαλίσουμε όλους τους αγοραστές Επίσης το roaming, η περιαγωγή εδώ δεν έχουμε εσωτερική αγορά, έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ κρατών και όχι μεταξύ εταιριών. Η δική σας στρατηγική ποια είναι σε σχέση με την περιαγωγή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο καθηγητής Κορέια Δεκάμπος. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος, γι' αυτό θα ήθελα να σας υποβάλω μια πρόταση. σε σχέση με την νομοθετική διάχυση. Σας προτείνω να αλλάξουμε τρία προγενέστερα έργα με ένα καινούριο. Δηλαδή κάθε φορά που προβάλλεται μια νέα νομοθετική πρόταση θα πρέπει να ψάξετε στον κατάλογο της νομοθεσίας για να δείτε ποια είναι τα δύο ή τρία έργα τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν το νέο έτσι ώστε να μπορέσουμε με κριτικό μάτι να δούμε την παλαιά νομοθεσία και επίσης να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις νέες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι αφήσατε την τελευταία πρόταση ε, ως καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί τηρήσατε το χρόνο. Ξέρω ότι ο Επίτροπος πρέπει να φύγει σχεδόν αμέσως, αλλά έχετε το λόγο, Μισελ Μπαρνιέ, για άλλα ε, ζητήματα τα οποία θίγησαν τώρα. Εντάχει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι αδειμονείτε να περάσετε στο επόμενο θέμα, στις σημαντικές ψηφοφορίες. Ο κύριος Δεκάμπος έκανε μια πολύ ευφυή πρόταση. Εγώ ήμουν βουλευτής 20 χρόνια στη χώρα μου και στη Γαλλία είδα ότι πάντα ψηφίζουμε νέους νόμους χωρίς να αποτιμούμε τους παλαιότερους ε, βεβαίως έχει μεγάλη σημασία να ε, είμαστε ιδιαίτερα εποπτικοί και να αναθεωρούμε οδηγίες. Δεν ξέρω κατά πόσο στο τομέα της εσωτερικής αγοράς υπάρχουν 1.400 έως 1.600 κείμενα τα οποία είναι αναθεωρήσιμα. Μερικά από αυτά είναι και άχρηστα. Εν πάση περιπτώσει μιλάτε για ένα προς τρία. Πολύ ψηλή αναλογία. Βεβαίω είμαι ε, ιδιαίτερα δύσπιστο και ως προ τα στατιστικά στοιχεία. Θα ήθελα όμως με διάβγεια να δούμε τα κείμενα τα οποία πια δεν είναι αποτελεσματικά ή δεν έχουν και χρησιμότητα. Ως προ τον κύριο Ζουβέ και την κυρία ε, Ράπτη έθιξαν την ελληνική κρίση Θα ήθελα να είμαι σαφής ως προς αυτό το ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό. Βεβαίως η Ελλάδα διανύει μια πολύ δύσκολη κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιήθηκε με βάση τη δέσμευση Μπαρόζο ολιρέν, Ρεν μαζί με την ΕΚΤ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου έτσι ώστε να σκιαγραφίσουν τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προαπαιτείται αυτή η αλληλεγγύη και θα πρέπει βεβαίως όλα αυτά να γίνουν μέσα στα πλαίσια μιας πειθαρχία. Η Ελλάδα ανέλαβε αυτή την πειθαρχία με μεγάλο θάρρος και καταλαβαίνω κυρία Ράπτη ότι το ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος είναι πολύ υψηλό. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι και οι άλλες χώρες είναι ε, έτοιμες να συνδράμουν. Κύριε Ζουβέ, κυρία Ράπτη, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μαθήματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή την κρίση για τη ζώνη του ευρώ για την ευρωζώνη χρειάζεται μια διαρκής οικονομική εποπτεία και συντονισμός και μια οικονομική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση δεν είναι πια μια μεγάλη λέξη, ποτέ δεν ήταν. Χρειάζεται πειθαρχία από όλους, γιατί όλοι προσυπογράφουμε το ίδιο συμβόλαιο. Θα πρέπει επίσης να έχουμε άμεμπτα στατιστικά συστήματα για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, γιατί ακριβώς μιλάμε, ακριβή αριθμητικά στοιχεία και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς και με τον συνάδελφο ΡΕΝ φτάνουμε στα, σε απτά αποτελέσματα και συμπεράσματα για ρύθμιση, για διαφάνεια της αγοράς σε όλες τις αγορές. Και γι' αυτό θα υποβάλω ένα σχέδιο στο Κοινοβούλιο το καλοκαίρι για την γενική ε, ρύθμιση των παραγόγων. Κύριε Μάντερς, γνωρίζω τις ε, δυσκολίες εφαρμογής οδηγιών. Νομίζω ότι ο μηχανισμός ε, της διευθέτησης είναι πάρα πολύ καλός. Τις ε, επόμενες εβδομάδες, με βάση τις διαβουλεύσεις, θα υποβάλω προτάσεις για το γλωσσικό καθεστώς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Υπό Ισπανική Προεδρία θα γίνει αυτό. Ως προς το θέμα του κατακαιρματισμού της εσωτερικής αγοράς και του πότε θα ανοίγουν και θα κλείνουν οι μεγάλες επιφάνειες, θα δούμε τα δίκτυα διανομής και τα δίκτυα λιανικής πώλησης και θα συμπεριλάβω σε αυτή την εργασία μία γενικότερη διάγνωση αυτού του κατακαιρματισμού της αγοράς, ιδιαίτερα σε περιόδους εκπτώσεων, προσφορών κλπ. Θα δούμε λοιπόν αυτό το θέμα της ε, ε, Λιανικής. Κύριε Κρές, έχετε αναλάβει μια πολύ δύσκολη έκθεση. Θα βρούμε τον τρόπο να ορίσουμε, να οριοθετήσουμε σωστά την εσωτερική αγορά. Αυτό είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί η έκθεση αυτή συνεισφέρει στον ανθρωποκεντρισμό αυτού του σχεδίου. Κυρία ε, Βερνιό, δέχομαι την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Χάρτα, την επαγγελματική κάρτα δηλαδή του καθενός τουλάχιστον για τα βασικά επαγγέλματα, μιλάμε για προστασία, αλλά όχι για προστατευτισμό. Δεν είμαι προστατευτικός, υπέρ του προστατευτισμού δηλαδή. Εάν δεν αποκομίσουμε όλα τα διδάγματα που πρέπει, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέες κρίσεις, διότι ο ρυθμός των αγορών είναι πολύ υψηλότερος από τον πολιτικό λόγο. Η αγορά υπέστη επίσης πλήγμα. Εάν δεν ε, αδράξουμε αυτά τα διδάγματα, τότε θα αντιμετωπίσουμε μια νέα κρίση στα πλαίσια της ενίας αγοράς. Διότι θα υπάρξουν ε, λαϊκιστικές αντιδράσεις προστατευτισμού και άρα η εσωτερική αγορά θα είναι το πρώτο θύμα. Θα εργαστώ λοιπόν κατά τους προσεχείς μήνες για την ε, πρόσβαση των ΜΜΕ στα χρηματιστήρια. Ε, κύριε Μπάντ, δώστε μου χρόνο για να έχω μία ε, διαυγή θέση ως προς την οδηγία πλαίσιο που θέλουν μερικοί, οδηγία ποιότητας, όπως είπε πρόεδρος Μπαρόζο, ένα νομοθετικό πλαίσιο με τομεακές οδηγίες των δημοσίων αγορών προμηθειών. Στόχος βεβαίως παραμένει η προστασία. Συνεργαζόμαστε με τους κυρίους Ταγιάννη και Κρές για να φτάσουμε σε μία ψηφιακή ευρωπαϊκή πολιτική, βιομηχανική πολιτική. Προς τον κύριο Βάντερ Κάμπ θα ήθελα να πω ότι θα σας κοινοποιήσω την ε, ανακοίνωσή μου για την εφαρμογή της οδηγίας περιπηρεσιών. Σας έδωσα ακριβή αριθμητικά στοιχεία για τον ρυθμό μεταφοράς από τα κράτη-μέλη. Έχουμε 600 εθνικά κείμενα τα οποία έχουν τροποποιηθεί, αλλά βρίσκεται σε καλό δρόμο η οδηγία, η μετάταξη της οδηγίας. Προς την κυρία Στήλερ, θα ήθελα να πω ότι θα συνεργαστώ με τον Επίτροπο Νταλή για την καταναλωτική πίστη. Προσπάθησα να προωθήσω την ιδέα του ένομου ε, δανείου. Θα πρέπει να ε, προστατεύουμε και τον δανειολήπτη και τον δανειοδότη και προσπαθώ να δώσω τελική μορφή στις διαβουλεύσεις για να δούμε τι επιλογές έχουμε μέσα στα πλαίσια των γενικών νομοθετημάτων. Mm-hmm. Κυρία Τούν, σας ευχαριστώ για την πρόταση του φόρουμ. Στην αρχή της Πολωνικής Προεδρίας θα πρέπει να λάβει χώρα αυτό το φόρουμ. Δεν λέω πού, δεν λέω πού. Λοιπόν, τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό και η Κομισιόν, καθώς και η κοινωνία των πολιτών, όλοι μας θα πρέπει να επεξηγήσουμε τα κείμενα, τους νόμους και να ενισχύσουμε αυτή την ανθρώπινη διάσταση. Στο πρώτο αυτό φόρουμ θα προβούμε σε ένα βαθμολόγιο, θα συντάξουμε ένα βαθμολόγιο για να δούμε πού βρισκόμαστε ως προς τις ενιαίες θηρίδες και τα αποτελέσματα του Solvit. Όλοι θα είναι στο επίκεντρο αυτού του φόρουμ εσωτερικής αγοράς που προτείνατε. Σας ευχαριστώ. Uh, um, Επίτροπε, αυτό το χειροκρότημα δείχνει πόσο αποδεκτή είναι η δέσμευσή σας και πόσο σας εκτιμούμε στην Επιτροπή μας. Πραγματικά έχετε εξαιρετική δουλειά κάνει και σας περιμένει και άλλη τόση. Ελπίζω ότι μπορώ να μιλήσω ονόματο όλων των μελών τη Επιτροπής μας. Ε, μακάρι να σα μοιάζαμε και στον ενθουσιασμό σα και στη δουλειά που κάνετε. Έχετε πολύ σαφεί στόχου για να λειτουργήσει καλύτερα η εσωτερική αγορά για του ε, πολίτε και για την προστασία των καταναλωτών και βεβαίω ε, θα σα βοηθήσουμε κι εμεί όσο μπορούμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και βεβαίω πάντα είσαστε ευπρόσδεκτοι στην Επιτροπή μας.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 Uh, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε γιατί πρέπει να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ καθίστε, επαναλαμβάνω, και κάντε και λίγη ησυχία για να ψηφίσουμε. Καταρχάς, να ελέγξουμε λίγο το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αν δουλεύει καλά. Θα το κάνουμε με τον συνηθισμένο τρόπο. Όλα τα μέλη του ΕΛΚ που θα ψηφίσουν, παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Όλα τα μέλη του ΕΛΚ που θα ψηφίσουν, ψηφίστε τώρα. Για να ελέγξουμε. Επαναλαμβάνω, το ΕΛΚ. Είναι ένας παραπάνω. Πρέπει να είναι 40. Α, η κυρία Βάιλερ ψήφισε. Η κυρία Βάιλερ ψήφισε για το ΕΛΚ. Προφανώς. Τέλο πάντων, κλείνουμε αυτή την ψηφοφορία, να ξαναρχίσουμε. Πέρα της ψηφοφορία. Λοιπόν, το ΕΛΚ μόνο παρακαλώ. Μόνο το ΕΛΚ θέλει να το ξαναελέγξουμε. Μόνο τα μέλη του ΕΛΚ, επαναλαμβάνω, ψηφίστε τώρα. Right, that's 14. 14 αυτή τη φορά, μάλιστα. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κυρία Βάλερ, τώρα μπορείτε να ψηφίσετε. Right, that's correct. We have Σωστό. 10. Φιλελεύθεροι. Oh, sorry, you've gone one over now. Oh, ένας παραπάνω είναι τώρα. Ξανά οι σοσιαλιστές. Όλα τα μέλη των σοσιαλιστών παρακαλώ ψηφίστε. 11. 12 τώρα. Πάλι από την αρχή πάμε. Να κλείσουμε αυτή την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Λοιπόν, πέρας ξανά οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Σοσιαλιστές και δημοκράτες μόνο παρακαλώ. Παρακαλώ ψηφίστε. Fine. So that's... Μπράβο. Πολύ ωραία. Πέρασε. Φιλελεύθεροι. Έναρξη ψηφοφορίας για τα μέλη των φιλελευθέρων. Τέσσερις. Πολύ καλά. πράσινη η πράσινη παρακαλώ. Τρίση. τρίση, Συντηρητικές και μεταρρυθμιστές. Τρεις. Γκουε. Δύο. Σωστά. Πολύ ωραία. Και δεν έχουμε ε, ελεύθερους δημοκράτες. Μάλιστα. Περνάμε στην ε, έκθεση της κυρίας Φάιλερ. Μήπως θέλετε να πείτε ορισμένα πράγματα πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που μετά από μια τόσο ταραχώδη ε, γνωμοδότηση καταφέρουμε να φτάσουμε σήμερα στην πρώτη ψηφοφορία. Να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτά που είπε ο Επίτροπος Μπαρνιά στη συζήτηση για το πόσο σημαντικές είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πόσο σημαντική είναι η δική μας βοήθεια για την εσωτερική αγορά και τις δυνατότητες που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομίζω ότι αυτή η νομοθετική πρόταση είναι πραγματικά ένα σημαντικός πυλώνας για τη βοήθεια αυτή. Και μετά από μεγάλες τρικυμίες καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό, όπως είπα στην γνωμοδότησή μου. Οι συμβαστικέ προτάσει πρέπει να, έχει, να είναι βρίσκονται μπροστά σα. Θα ήθελα να σα αναφέρω ποιε είναι οι πιο σημαντικέ. Η πρώτη είναι ότι έχουμε αλλάξει την ε, προθεσμία για τις, ε, για πληρωμές και την έχουμε κάνει 30 ε, ημέρες με ανοίγματα για τις δημόσιες υπηρεσίες τις επιχείρησεις μέχρι 60 ημέρες και με ένα παραθυράκι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με ένα παράθυρο. Επίσης υπάρχει το θέμα της ελευθερίας των μεμονωμένων συμβάσεων. Ε, δεν έχουμε το αρχικό στάτους που ήθελα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε προχωρήσει αρκετά και ως προς αυτό. Το δεύτερο, ο δεύτερος μεγάλος συμβασμός ήταν η διαγραφή του 5% των κυρώσεων για, την, για το δημόσιο τομέα. Η πρόταση αυτή από την Κομισιόν από την αρχή ήταν αμφιλεγόμενη. Ευχαριστώ το Άλντε που αυτό, αυτή την ποινή του 5 7% δέχτηκε να αλλάξει ε, και δέχτηκε να συμφωνήσει με τον ε, συμβιβασμό μας. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν οι, οι φορείς τι γίνεται και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Το 5% έχει διαγραφεί, λοιπόν. Τρίτο σημείο για τα recovery costs έχουμε ένα αρκετά απλό σύστημα. Μια, ένα συνολικό ποσό χωρίς περίπλοκα, χωρίς περίπλοκα ποσοστά 40 ευρώ. Ε, χαίρομαι που συμφώνησαν οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι αυτός είναι και πιο εύκολος τρόπος. Ε, τέταρτο επαλήθευση για τις μέχρι 30 ημέρες για μεγάλες κατασκευές, για μεγάλες εγκαταστάσεις. Ε, θα ήθελα εδώ να σας πω ότι μέχρι 30 ημέρες είναι το όριο. Φυσικά μπορεί να είναι και πιο μικρό. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε και τις 30 ημέρες. Και τελευταίο σημείο, τα επιτόκια. πρώτα στις Κομισιόν 7%. Εμείς συμφωνήσαμε να πάνε να αυξήσουμε κατά 2% και να πάμε στο 9%. Νομίζω ότι είναι πιο πρακτικό και πιο λογικό. Είναι σημαντικό ότι ισχύει και για δημόσιε επιχειρήσει και για ε, ιδιωτικέ. Ε, λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη μα την επιθυμία του Κοινοβουλίου να υπάρχει δηλαδή η συμμεταχείριση και για του δύο, και για τον ιδιωτικό και για τον δημόσιο τομέα. Και αυτό ο κανόνα ισχύει και ε, εφαρμόζεται και στις ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις και στις δημόσιες. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Ίσως ε, να υπάρξει κάποια ακόμη τροπολογία για ένα σημείο το οποίο υποστηρίζω εγώ βέβαια. Θα το δούμε, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα τα χρονικά, τη χρονική μας οργάνωση, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να προετοιμάσουμε και τελεσίδικα την, την κατηγορία α, ψηφοφοριών, δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε το τελευταίο σημείο. Τώρα, κάποια θέματα που δεν θα βρείτε στο συμβασμό είναι γιατί, όχι γιατί διαφωνήσαμε, αλλά γιατί θεωρήσαμε ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να καταλήξει στη θέση της για την πληροφορία, δηλαδή η συμπερίληψη της οδηγίας 17, καθώς επίσης η ίδια μεταχείριση και για τα νοσοκομεία. Ε, ελπίζω να λάβουμε μεγάλη ε, πλειοψηφία. Και επίσης να ευχαριστήσω την Κομισιόν η οποία έδειξε τεράστια ευελιξία γιατί με την πρόταση αυτή και με τον συμβασμό και με τις ε, συμβαστικές τροπολογίες σίγουρα για κάποια ε, σημεία πιέσαμε την Κομισιόν. Γιατί πραγματικά φέραμε τα πάνω κάτω στην πρότασή της και παρόλα αυτά η Κομισιόν δούλεψε πολύ επικοδομητικά και συνεργάστηκε ώστε να καταλήξουμε σε κάτι ε, που να μας ικανοποιεί και τους δύο. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ ηγηθήκατε αυτή τη διαδικασία ε, πολύ αποτελεσματικά. Χαίρομαι που καταλήξαμε στο κείμενο αυτό. Ευχαριστώ και όλη την, ε, όλο το προσωπικό που προετοίμασε τι ε, τις ε, ε, λίστες ψηφοφορίας, τους καταλόγους γιατί πραγματικά περάσανε πολλέ ώρε το βράδυ εδώ. Λοιπόν, πάμε στην τροπολογία 54 ε, για το άρθρο 1. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε. Άρθρο 2. Ορισμοί. Υπάρχει ένα μπλοκ ε, από τον κύριο Μάντερ, 55-67, ε, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Ο κύριος Μπουζόη, 56, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τρεις ίδιες, Σαλβίνη Μπαρτολότσι Πιτέλα, υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Πάμε. Άρθρο 2.2. Τροπολογία 6 της κυρίας Βάιλερ, της συγγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 6, σημείο 2, τμήμα 2 από την κυρία Βάιλερ. Υπέρ. Κατά. Για πάλι. Νομίζω ηλεκτρονικά να το δούμε αυτό καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την τροπολογία 6 τμήμα 2 της κυρίας Βάιλερ. Vote is open. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 21 έναντι 15 ψήφων υπέρ. Πάμε στην 6-3 της κυρίας Βάιλερ. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 υπέρ 21 κατά. Τροπολογίες από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Ναι, αλλά απορρίφθηκε. Μήπως πρέπει να ψηφίσουμε γι' αυτό. Όχι, εντάξει. Νομίζω καλύπτονται και κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο σημείο. Απορρίπτεται το 63, οπότε έχουμε τώρα ένα μπλοκ τροπολογίων 62, 63, 65. Επιτροπή Βιομηχανίας, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 64 αποσύρεται από την, Κυριακό, από την κυρία Κόμη, της ε, κυρίας Ροϊτόβα 66 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε, ούτε της κυρίας Χάντσλικ. 68, πάμε στην 69 του κυρίου Αρία Σετσοβερία. Υπέρ. Πάμε στην ε, κατευθείαν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. 69, τροπολογία 69 του κυρίου Τσιβερία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 20 προς 15. Πάμε στην πρώτη συμβαστική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 78, 79, 146, 147. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Πάμε σε δύο από τον κύριο, από τον κύριο Κρόιτσμαν. Α, όχι. Πάμε στη συμβαστική πρόταση 2. Συγγνώμη, συγγνώμη. Γιατί είδαμε τις άλλες 4. Λοιπόν, τροποποιητική, ε, συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται από τη συμβαστική 2, συγγνώμη, πάμε στην συμβαστική 3. Άρθρο 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε. Πάμε στην τροπολογία 87 του κυρίου Μάντερς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η Γιούρι 7 καταπίπτει. Α, όχι, συγγνώμη. Πρέπει να ψηφίσουμε την 7 της, ε, νομικών υποθέ... της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 4. Αλλά έχουμε χωριστή ψηφοφορία, ψηφοφορία κατά τμήματα. Ας το πάρουμε λοιπόν όπω είναι και στο κείμενο. Ας δούμε το πρώτο τμήμα για το 2α και το πρώτο τμήμα του 2β μέχρι το 60 ημέρες. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και πάμε στο τμήμα 2. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Δεν λέει ότι υπάρχει τροπολογία προφορική εδώ. Η κυρία Χάνσλεκ θέλει να προτείνει κάτι. I have here, but I think you need to read You have, you... Έχετε λάβει την ε, προφορική μου τροπολογία και γραπτός. Λοιπόν, εναλλακτική σε αυτό που υπάρχει στην, ε, στον κατάλογο ψηφοφοριών. Μάλιστα. Να το διαβάσω. Λοιπόν, ψηφίσαμε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η προθεσμία πληρωμών που υπάρχει στην σύμβαση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 60 μέρες. Ε, αυτό το ψηφίσαμε. Και τώρα η αναδιατύπωση λέει ότι θα πρέπει να, συμφωνήσουν, να συμφωνήσει ο πιστωτή ε, ε, σύμφωνα, ε, εφόσον η, κάποια, η συμφωνία αυτή δεν είναι επιζήμια προς κάποιο από τα συμβαλόμενα μέρη. Η κυρία Βάιλερ. μια ασάφεια επικρατεί. Η διατύπωση, η πρώην προηγούμενη διατύπωση λέει για unjustified damages τι ε, ζημιές ζημιέ. Την είχα επικρίνει γιατί είπα ότι είναι ασαφή. Τώρα που λέει not grossly unfair, που δεν είναι ιδιαζόντω άδικη, ε, νομίζω ότι είναι καλύτερη και θα την υποστηρίξω. Να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Θέλετε κάτι διαδικαστικό. Έχω το λόγο. Όχι. Πες μου τι θες να πεις και θα δούμε. Για την προφορική τροπολογία, Πρόεδρε. Και γιατί να μην τη βάλουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να μιλήσω. Μιλήστε. Ευχαριστώ. Η αρχική πρόταση του ΕΛΚ για την προφορική τροπολογία περιλάμβανε και να αλλάξει στο ακτιμώντα, στην ανατολική σκέψη, και αυτό το κομμάτι που έλεγε για τις 60 μέρες. Μήπως είναι δυνατόν, συνάδελφοι, να μείνουμε σε αυτό που είχαμε στην αρχική πρόταση, που θα λέει το εξή. Σύμφωνα, ε, ακολουθώ οι συμφωνίε που γίνονται για τι προθεσμίε πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων θα πρέπει να, ε, να ακολουθούν τι 60 ημέρε αντί να περιορίζονται. Το γενικό κανόνα των 60 ημερών δηλαδή. Για την ελευθερία των συμβάσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, ναι, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα που λέτε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το δεχτούμε τώρα αυτό. Εγώ τώρα έχω μπλεχτεί τελείω. Δεν ξέρω τι ακριβώ θέλετε. Η κυρία Χάνσλικ έχει υποβάλει ε, εκ μέρου του ΕΛΚ προφορική τροπολογία, την οποία δέχεται η συγγήτρια. Οπότε να την ψηφίσουμε. Ε, ε Α είμαστε και λίγο πειθαρχημένοι, έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε ο καθένα ό,τι θέλει τώρα. Well, let me just clarify, because I think we do need... Λοιπόν, ε, πρέπει να προχωρήσουμε. Η κυρία Χάνσλικ προτείνει την προφορική της τροπολογία και το δεύτερο κομμάτι του 2β που σας διάβασα. Η κυρία Βάιλερ λέει ότι το δέχεται την διατύπωση αυτή. Οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Προφορική τροπολογία. Κυρία Κέπχαρτ. Πρόεδρε, ξέρω ότι η συγκήτρια διαφωνεί μαζί μου, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα το πω αυτό που θέλω, γιατί έχω την εντύπωση, έτσι όπως βλέπω τους ε, συναδέλφους μου, ότι υπάρχει μια σάφια. Ε, εμείς δεν δεχόμαστε να υπάρξει κι άλλη προφορική τροπολογία, να συμφωνήσει μεταξύ του το ΕΛΚ και να, να υποβάλει τις ε, τροπολογίες του στην Ολομέλεια. Αλλά τώρα θα ψηφίσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Αν θέλετε μετά να το συζητήσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Έτσι τώρα με ε, τροπολογίες που έρχονται και φεύγουν δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, αν οι ε, σοσιαλιστές απορρίψουν τροπολογία, εντάξει. Οπότε, ψηφίζουμε το υπάρχον δεύτερο τμήμα του κειμένου, γιατί μόνο αυτό μας έχει μείνει. Λοιπόν, το υπάρχον κείμενο το ψηφίζουμε τώρα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ωραία. Οπότε, συμφωνήστε με τις προφορικές τροπολογίες που θα κάνετε για να πάμε παρακάτω. Τώρα. Τροπολογία 96 της κυρίας Ρούιλε, 97 του Κρόιτσμαν και της Επιτροπής Βιομηχανίας. Είστε στη σωστή σελίδα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 96, το συγκεκριμένο τμήμα από την κυρία Ρούιλε, άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Uh, that is carried by 22 votes. Εγκρίνεται. συγγνώμη, 22 προς 13. Πάμε στην τροπολογία 6 από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Και αυτή να την ψηφίσουμε. Άρθρο 3, παράγραφος 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 3 καταπίπτει λόγω της συμβαστικής πρότασης και το 98 και 98. 101-102 καλύπτονται από το 4α αργότερα, οπότε πάμε στη συμβιβαστική πρόταση 5, σωστά? Πολύ ωραία. Συμβαστική πρόταση 5, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 104 του κυρίου Σαλβίνη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Πάμε στην 105 του κυρίου Πιτέλα και άλλων παρόμοιες ε, ταυτόσιμες ε, τροπολογίες υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 105 Πιτέλα και βιομηχανία υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην 105 το συγκεκριμένο τμήμα 3. Πιτέλα και Επιτροπή Βιομηχανίας υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Πάμε. Γιατί καταπίπτουν αρκετές τροπολογίες μετά από αυτές τις, ε, τις υπόλοιπες που πέρασαν. Πάμε στην παράγραφο 1. Τροπολογία Σαλβίνη. Σωστά. Όχι. It's going to be voted later, right, sorry. Okay. 121. 121, συγγνώμη. 121. 121 της κυρίας Ρόιτοβα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 125. Πάμε στην 128. 128. Της κυρίας Κόμη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 124 του κυρίου Αρεάς. υπέρ κατά απορρίπτεται 131 του κυρίου Μάγερ υπέρ πρέπει να ψηφίσουμε νομίζω ηλεκτρονικά 131 τροπολογία 131 του κυρίου Μάγερ ε, άρχεται η ψηφοφορία The vote is closed. That is carried. Ευχαριστώ. Πέρας ψηφοφορίας περνάει με 21 προς 15. Τροπολογία 8 της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 6. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, συμβιβαστική τροπολογία 7. Πε, ε, καταπίπτουν πολλέ τροπολογίε, πολύ καλή δουλειά τη εισηγήτρια. Συμβιβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 138. Η 145 και 144. Υπέρ, κατά. «138, 144, 145. Υπέρ. Α, έρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. The vote is Πέρας Απορρίπτεται. 13 προς 22. Πάμε στην 139 του κυρίου Μπουζόη. 139. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται 19 προς 17. Πάμε στην 142, Μάντερς. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θα προσπεράσουμε αρκετέ σελίδε τώρα γιατί καταπίπτουν διάφορε τροπολογίε και φτάνουμε στην 147, σημείο 3 τη κυρία Ρούιλε και της, των Επιτροπών Βιομηχανία Οικονομικών Υποθέσεων. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 147 τμήμα 4 της κυρίας Ρούλε υπέρ ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε καλύτερα 147 τμήμα 4 της κυρίας Ρούλε άρχεται η ψηφοφορία The vote is closed. Uh, that is... Απορρίπτεται 16 προς 19 Πάμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Τροπολογία 9, τμήμα 1. Υπέρ κατά εγκρίνεται του κυρίου Κάρας 150 υπέρ κατά εγκρίνεται βιομηχανία 9 162 υπέρ κατά εγκρίνεται 151 υπέρ κατά εγκρίνεται η 9 καταπίπτη. Προσπερνάμε και άλλες σελίδες τώρα. Πάμε στην 158, τμήμα 2, του κυρίου Κάρας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Στάιλερ. 172. Θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. 172 ε, τροπολογία της κυρίας Στήλερ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 προς 18. Πάμε. Πάμε στην 193 του κυρίου Πιτέλ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 194 του κυρίου Κρόιτσμαν. Υπέρ κατά απορρίπτεται. Πάμε στο άρθρο 6. Έχουμε παρόμοιες προπολογίες ε, από Ήτρα, Γιούρι, υπέρ, κατά. Περνάνε, εγκρίθηκαν. Μετά έχουμε μία σειρά σημείων, από των οποίων δεν θα ψηφίσουμε, εξαιτίας του ε, 150. Άρα θα πάμε απευθεία στην τελική έκθεση. Άρα τώρα πάμε στην 15. Σαβίνη. Άρθρο 7, παράγραφος 1. Υπέρ, κατά, καρνάει. 206, Σολβίνη. Καταπίπτει. Άρα είμαστε στο 7 παράγραφος 1α νέα. 13 και 14 Βάιλερ που ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ε, εγκρίθηκαν. Τροπολογία Ζουβέν που θα είναι προσθήκη στις 13 και 14 υπέρ των προσθήκων κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Άρα Ιουρί 15 και Ήτρε 16 καταπίπτουν. Άρθρο 7α νέο. 15 Βάιλερ υπέρ. Κατά εγκρίνεται 208 Χάντσλικ υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τώρα περνάμε σε ορισμένα άρθρα ε, Ιουρί 209 Σαλβίνη υπέρ κατά απορρίπτεται 210 Σαλβίνη υπέρ κατά απορρίπτεται πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις 7 16 Μότι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 υπέρ κατά απορρίπτεται 19 υπέρ κατά απορρίπτεται ε, το επόμενο μπλοκ η επόμενη σειρά σχετίζεται με προγενέστερες 23 λοιπόν που είναι προσθήκη του Γιούρι 1 αρχίζει η ψηφοφορία της ε, τροπολογίας κυρίας Κοράτσα Μπίλτ 23. The vote is That is carried by 20. Εγκρίνεται με 23 έναντι 10. Περνάμε τώρα σε μία σειρά τροπολογιών που δεν ε, ψηφίζονται διότι καλύπτονται ήδη, άρα τώρα περνάμε στο 18α νέο με την 51. Ιντάλγο Μούνι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Βάιλερ. 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5 Βάιλερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Μετά πάμε στην τελική ψηφοφορία. Έτσι δεν είναι κυρία Βάιλερ. Θα αρχίζει η ψηφοφορία, στη ψηφοφορία επί της τελικής πρότασης, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία ως προς την ε, τελική ψηφοφορία του κειμένου στο σύνολό του. Πέρασε. 30 υπέρ, καμία κατά και 6 αποχές. Σας ευχαριστώ. So, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βάιλερ. Θέλετε να πείτε λίγα λόγια. ησυχία, η συγγήτρια έχει το λόγο. Στο τέλος της πληροφορίας θέλω να τα πω, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την Γραμματεία της Επιτροπής και τους νομικούς συμβούλους μας και τους συνεργάτες βεβαίως όλων, γιατί πραγματικά έκαναν εξαιρετική δουλειά ε, θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Στην αρχή δεν το είχαμε προβλέψει ότι θα δουλεύαμε τόσο καλά μαζί. Και τέλο, να πω μια λέξη και για το Συμβούλιο. Βλέπετε μέσω τη σαφού ψηφοφορία και των σαφών πλειοψηφιών πώ γίνεται η δουλειά, οπότε πρέπει και εσεί να κινηθείτε. Ε, thank you very much indeed. Ευχαριστούμε κυρία Βάιλερ για αυτή τη δύσκολη ψηφοφορία και γιατί συνεργαστήκατε με τις Επιτροπές Νομικών Υποθέσεων και Βιομηχανίας. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Σας παρακαλώ όσοι επιθυμείτε να αποχωρήσετε χωρίς περιττές συζητήσεις, γιατί τώρα πρέπει να δούμε την επόμενη οδηγία για τα βιοκτώνα. Θέλετε το λόγο. Please, can you leave quietly? Thank you. Mrs. Sartori, do you want... Η κυρία Σαρτόρη, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση κανονισμού θέτει ως στόχο να αντιμετωπίσουμε το θέμα των βιοκτώνων έτσι ώστε η Οδηγία 98 να μετατραπεί σε ε, κανονισμό. Έγινε μια συζήτηση στην Επιτροπή Βιομηχανίας μαζί με τους ε, σκιώδεις και ελπίζω να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το ζήτημα με μια ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να τονίσω στους συναδέλφους ότι αυτή είναι μια γνωμοδότηση ε, όπου συνεργαστήκαμε με ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή Βιομηχανίας. Άρα η ενισχυμένη συνεργασία ε, είναι αποτελεσματική. Έκθεση Σαρτόρη, άρθρο 1, παράγραφος ε, ε, τροπολογία 4. That Εγκρίνεται. 5. Σαρτόρι. Υπέρ. That. Κατά. Νομίζω θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρθρο 5. Σαρτόρι. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Uh, that is uh, that is carried. Περνάει 23 υπέρ 9 κατά. 108 Γκέπχαρτ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 109 Φόξ Βάις Γκέρμπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 Σαρτόρι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 110 αρχίζει η ψηφοφορία για την 110. Σαρτόρι. Πέρας. Εγκρίνεται με 23 έναντι 13 ψήφων. 7. Σαρτόρι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 110 σχετίζεται με την 109, 8 σαρτόρι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 9 σαρτόρι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 10 σαρτόρι υπέρ, κατά, επίσης εγκρίνεται. 11 σαρτόρι υπέρ, κατά, εγκρίνεται άρθρο 4, παράγραφος 1, 12 ε, της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. Άρθρο 5 τώρα, 14 σαρτόρι υπέρ, μάλλον ε, άρχεται η ψηφοφορία, 14 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, το ΕΛΚ έχει συν 2, επιπροσθέτως 2. Ας ξαναγίνει η ψηφοφορία. Έλεγχος παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία εκ νέου. Ελπίζω να έχουμε το σωστό αριθμό από το ΕΛΚ. πέρας 23 έναντι 13. Ωραία. Ε, Μπουζόη 112 καταπίπτει 15 σαρτόρι. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 15 σαρτόρι. πέρας εγκρίνεται με 21 ψήφους έναντι 13. 16 Σαρτόρι. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 16. Ε, The vote closed. Πέρας εγκρίνεται με 26 υπέρ 10 κατά. 17 Σαρτόρι. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 17. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 έναντι 13. Άρθρο 7. 113 Κέπχαρτ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 113. Πέρας. 31 ψήφι εναντί 2. 18 Σαρτόρι. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. That is carried by 31. ψήφοι υπέρ, 4 κατά. 19 σαρτών. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. That is carried by 23. Περνάει με 23 έναντι 11. 20 σαρτόρι. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται 22 έναντι 13. 21. 21. Σαρτόρι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 8. Τροπολογία 22. Σαρτόρι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 23. Σαρτόρι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 9. Παράγραφος 24. Σαρτόρι, η, μάλλον άρχεται η ψηφοφορία για την 24. Πέρας εγκρίνεται. 20 υπέρ έναντι 13. Κατά. Άρθρο 10, παράγραφος 3, τροπολογία 114 με μια προφορική Κέπχαρτ που φαίνεται στον κατάλογό σας υπέρ κατά εγκρίνεται. Άρα εκπίπτει η επόμενη. Λοιπόν, 25 άρθρο 12 σαρτόρι υπέρ κατά εγκρίνεται. Άρθρο 15, τροπολογία 115, μπουσόι. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed πέρας. Εγκρίνεται με 21 ψήφους εναντί 13. 26. Σαρτόρι. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 26. Σαρτόρι. Πέρας. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ 15 κατά. 27. Σαρτόρι. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται 22 έναντι 13. Τώρα, περνάμε στις προφορικές τροπολογίες Fox Artori, Μπουζόη. Άρθρο 15, παράγραφος 5. Υπέρ, παρακαλώ, κατά. Εγκρίνονται. Άρα, τώρα περνάμε στην 29, Σαρτόρι. Υπέρ, κατά εγκρίνεται 30 σαρτόρι υπέρ κατά εγκρίνεται 31 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 22 υπέρ 13, 13 κατά 32 σαρτόρι υπέρ κατά Εγκρίνεται. Άρθρο 17. Τροπολογία 116. Μπουσόη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 117. Μπουσόη. Υπέρ. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε. Μάλλον υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 118 μπουσόι υπέρ κατά απορρίπτεται 119 μπουσόι με μία προφορική που φαίνεται στον κατάλογο υπέρ κατά εγκρίνεται Κριστιαν πέρασε και μία δική σου τα κατάφερες άρα 119 κατά πίπτη άρθρο 18 Έχουμε μία ενοποιημένη τροπολογία Σαρτόρι Μπουσόι σε δύο τμήματα που φαίνονται στον καταλογό σας ποιοι είναι υπέρ του τμήματος 1 της ενοποιημένης. Κατά εγκρίνεται και τώρα το 2 ψηφίζουμε, το τμήμα 2. Ποιοι είναι υπέρ του τμήματος 2. Κατά επίσης εγκρίνεται. Άρα μετά την ενοποιημένη υπάρχει μια σειρά που καταπίπτουν 34 σαρτόρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 σαρτόρι υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά εγκρίνεται. 37 υπέρ όχι Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 37. Ε, Πέρας. Εγκρίνεται με 22 εναντί 13. 38. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 38. Πέρας. 22 έναντι 13. Εγκρίνεται. 39. Σαρτόρι. Αρχίζει η ψηφοφορία. 39. Πέρας. Περνάει 19 έναντι 15. 40. Σαρτόρι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 41. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 41. Πέρας. 23 υπέρ, 12 κατά. Τώρα προχωράμε, ψηφίζουμε τη, επί του 21, του άρθρου 21. Όχι, γιατί απορρίφθηκαν οι προηγούμενες 44 σαρτόρι. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 44. Uh, the vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται 22 1 13. Άρα η 122 μπουσόι που είναι προστήκη δύο λέξεων, ποιοι είναι υπέρ της προστίκης αυτής, κατά, εγκρίνεται. Άρθρο 22, Εσίος, 45, Γκέπχαρτ, με την προφορική τροπολογία που βλέπετε στον κατάλογο. Ποιοι είναι υπέρ της 45 με την προφορική κατά, εγκρίνεται. Σε αυτή την περίπτωση, λέει ο πρόεδρος και διακόπτη, καταπίπτουν όλες οι υπόλοιπες. Πάμε στις 46 λοιπόν ψηφίζουμε την 46 Σαρτόρι. 46-47 μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται. 48 Σαρτόρι υπέρ παρακαλώ. Ψηφίζει το ΕΛΚ. Κατά. Δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, 48. Ε, ΕΛΚ, συγκροτηθείτε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. 50. Σαρτόρι. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 50. The vote is closed. Πέρασε, περνάει 22 εναντί 13. 51. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 51. That is carried. Πέρασε 23 εναντί 13. Άρθρο 25 εσίως. Κοινή, μάλλον συναρμοδιότητα εδώ. 52 Σαρτόρι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 27. 53 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 28. Τροπολογία 123. Γκέπχαρτ. Αρχίζει η ψυχοφορία επί της 123. The vote is closed. Uh, that is defeated by 20. Απορρίπτεται 20 κατά. Άρα έχουμε την 55 σαρτόρι υπέρ κατά εγκρίνεται 56 υπέρ κατά εγκρίνεται 57 υπέρ κατά εγκρίνεται Άρθρο 29, 58 Σαρτόρι υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 59 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρθρο 33, τροπολογία 124, Κρόιτσμαν, υπέρ, μάλλον αρχίζει η ψηφοφορία, ονομαστική, επί της 124, Πέρας απορρίπτεται 19 κατά 17 υπέρ. 125 μπουσόι. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 126 φόξ σαρτόρι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται άρθρο 33α, νέο άρθρο. Έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία σε τρία, μάλλον όχι, σε δύο τμήματα, γιατί το δεύτερο, το αρχικό δεύτερο έχει αποσυρθεί. Άρα ψηφίζουμε το 127 τμήμα 1, όπως φαίνεται στον καταλογό σας, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα, το δεύτερο το αρχικό έχει αποσυρθεί, Άρα ψηφίζουμε το 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 60. Σαρτόρι. Ψηφίζουμε την 60 ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Για την 60 πέρας εγκρίνεται 21 ψήφοι εναντί 12. 61. Ε, σαρτόρι Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. 23 έναντι 10. 62. Σαρτόρι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 129. Μπουσόι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 63. Σαρτόρι υπέρ κατά εγκρίνεται. 40, 64. Ενισχυμένη συνεργασία. 64 ε, και 130. Σαρτόρι Μπουσό υπέρ κατά εγκρίνονται. Άρθρο 44 παράγραφος 3. 65 υπέρ Α, καλύτερα να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. 65 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 26 προς 9 εγκρίνεται. Περνάμε στην 131, που καταπίπτει βέβαια. Οπότε πάμε στην 66. Σαρτόρι, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. 67, Σαρτόρι. Άρχεται η ψηφοφορία για την 67. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται 25 προς 9. Και τώρα περνάμε στο άρθρο 46, ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Τεσσάρων πολιτικών ομάδων, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε, πάμε στην 136 του κυρίου Μπουσόη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Τριών πολιτικών ομάδων. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 προς 12. 76 στο άρθρο 48. 76. Υπέρ. Έναρξη ψηφοφορίας. The Εγκρίνεται 23 προς 13. 13. 77 της κυρίας Σαρτόρη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 78 Σαρτόρη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 49. 79. Σαρτόρι. Έναρξη ψηφοφορίας. Μιλάμε για το άρθρο 49, τροπολογία 79 της κυρίας Σαρτόρι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 22 προς 13. Τροπολογία 80 Σαρτόρι. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 22 προς 12. Τροπολογία 81. Άρθρο 52. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 53. Τροπολογία 82. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 82. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 προς 12. 54, τροπολογία 83 Σαρτόρι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 143 Εύλιν Γκέπχαρτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 144 Γκέπχαρτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 145 Γκέπχαρτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 146 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για, το για την 146. The vote is closed. Εγκρίνεται, ε, συγγνώμη, απορρίπτεται 18 προς 14, 147, Γκέπχαρτ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 84, Σαρτόρι ως προσθήκη, υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Περνάμε στο άρθρο 55. 85 σαρτόρι. Υπέρ. Κατά. Να ξαναρχίσουμε. Τροπολογία 85 σαρτόρι. Καλύτερα ηλεκτρονικός να ψηφίσουμε. Τροπολογία 85. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 προς 13. Τροπολογία 86 Σαρτόρι. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 22 προς 13. Τροπολογία 87. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 20 προς 13, 88 υπέρ. Εγκρίνεται 22 προς 13. 13. Περνάμε τώρα στο άρθρο 58, τροπολογία 89 της Αρτόρη. Έναρξη ψηφοφορίας για την 89. Πέρας. Εγκρίνεται 23 προς 13. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην προφορική τροπολογία 2 της κυρίας Σαρτορή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται επίσης. Περνάμε στο άρθρο 59. Τροπολογία 92 Σαρτορή. Τρία τμήματα. Ψηφίζουμε τώρα το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Συγγνώμη, μου είπαν ότι το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Γιατί εγκρίναμε την τροπολογία 85. Άρα χρειαζόμαστε κατά τμήματα ψηφοφορία ή όχι, Ρωτάω ο πρόεδρος. Δεν ξέρω. Προσπαθούμε να το ελέγξουμε. Σύμφωνα με τον κατάλογο ψηφοφορίας, ψηφίζουμε το άρθρο 59, παράγραφος 1α νέο. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Γιατί εγκρίναμε την 85. Θα το ψηφίζαμε μόνο αν είχε απορριφθεί η 85, αλλά η 85 εγκρίθηκε. Συμφωνείτε? Άρα δεν χρειαζόμαστε κατά τμήματα ψηφοφορία. Μπορούμε να ψηφίσουμε ολόκληρη την 92. Να ψηφίσουμε όλη την 92 λοιπόν. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στο άρθρο 62, τροπολογία 93 Σαρτόρι. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για το 93. Πέρας. Εγκρίνεται 23-13. 94. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 21 14. 95. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στο άρθρο 77, τροπολογία 148 του κυρίου Μπούσο, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 96. Σαρτόρι. Έναρξη ψηφοφορία για την τροπολογία 96. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 25 προ 8. Τροπολογία 149 Σαρτόρι. Έναρξη ψηφοφορία για την 149. Πέρας εγκρίνεται 23 προς 13. Τροπολογία 97 έχει αποσυρθεί, οπότε περνάμε στο άρθρο 81, τροπολογία 98. Υπέρ της 98, κατά, εγκρίνεται. 150-151 μαζί τις ψηφίζουμε. Έναρξη ψηφοφορίας για τις τροπολογίες 150 και 151. Πέρας. Είχαμε έναν παραπάνω. Μήπως να το ελέγξουμε. 23-14. 23-13 μάλλον, γιατί ένα ήταν παραπάνω. Άρθρο 82, 152, Fox και Weisberger, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Άρθρο 83, τροπολογία 99, Σαρτόρι, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 100, Σαρτόρι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται επίσης. Τροπολογία 153, Μπουζόι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 154. Μακλάρκιν και Μπουζόι. Έναρξη ψηφοφορίας για την 154. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 26 προς 10. Περνάμε τώρα στα εκτιμώντας. 11α νέο, προφορική τροπολογία, σαρτόρι, μπουσόι και φόξ, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 101. Δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε γιατί νομίζω ότι θεωρείται ότι εγκρίνεται ή απορρίφθηκε ανάλογα με, τις με τη προηγούμενη ψηφοφορία. Οπότε, περνάμε, νομίζω, στην τελική ψηφοφορία τώρα. Τελική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας ε, για την ε, έκθεση. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 προς 3. Εννέα αποχέ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σαρτόρη. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας δουλειά και περιμένουμε τα αποτελέσματα στην Επιτροπή περιβάλλοντο. Συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο. Έχουμε τη γνωμοδότηση του κυρίου Μπουτσόη για τα ιατρικά προϊόντα και δίνω το λόγο στον εισηγητή. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο γνωμοδότησης που θα ψηφίσουμε είναι το αποτέλεσμα μηνών εργασίας, ε, συνεργασίας ε, με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, ε, στα οποία είμαι ευγνώμονες. Οι τροπολογίες βελτιώνουν το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όταν λέω βελτιώνουν εννοώ από πλευράς ασθενών. Θα θέλαμε να κάνουμε δύο σύντομα σχόλια. Πρώτον, θα ήθελα να διευκρινίσω το γεγονός ε, ότι θα ήθελα να υποστηρίξω τη συμβιβαστική 1 παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται αυτό στον κατάλογο ψηφοφορίας. Είναι ένα σφάλμα. Και επίσης προφορική τροπολογία στο άρθρο ε, β ε, νέο και έχετε και το νέο κείμενο στη διάθεσή σας και θα το ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίστιαν. Οπότε να περάσουμε στην ψηφοφορία ευθύ αμέσω. Τροπολογία 37. Βάι Χέμπερ και Μπουσό. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 38. Δεκάμπος. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορία από αυτού για την τροπολογία 38. Πέρας. Εγκρίνεται 22 προς 12. Τροπολογία 3. Μπουσόι. Έτοιμα κατά τμήματα ψηφοφορίας. Πρώτο τμήμα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα τη τροπολογία 3, έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 προ 9. Μία αποχή. Δεύτερο τμήμα της τροπολογία. υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39, Ζουβέν και Βάις Γκέμπερ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 42 κάμπος, Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 43 ως προστίκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 41 καταπίπτει. 44. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. 6 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Το ψηφίζουμε ξεχωριστά. Έναρξη ψηφοφορίας. Ηλεκτρονικός. Μόνο για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας αυτής. Έχουμε ένα παραπάνω. Παρακαλώ αυτός που ψηφίζει δύο φορέ να μην το κάνει. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 24 προς 12. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Νομίζω χρειαζόμαστε ηλεκτρονική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 7. Ε, Πέρας. Εγκρίνεται 23 προς 13. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 45 καταπίπτει. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έχουμε συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα, περνάμε στην τροπολογία 51 Vice Geber Fox. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 9 καταπίπτη, Η τροπολογία 10 μπουζό υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 53 του κυρίου Μπουσόη. Ε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα 52-53 καταπίπτουν. Πηγαίνουμε στην 54 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 11. Καταπίπτει. 56. Μπουσόη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57 καταπίπτει. 12. Καταπίπτει επίσης. Τροπολογία 55. Του κυρίου Κορέα Κάμπος. Προστίκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Μπουζό υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ζιβέ Βαϊσμπέργκερ, τροπολογία 58 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ως προσθήκη. Τροπολογία 59. Κορέα Ντε Κάμπος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14 καταπίπτη. 60. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ έναρξη ψηφοφορίας ηλεκτρονικής για την 17. Πέρας. Εγκρίνεται 26 προς 10. 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κυρίου Ζουβά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορία για την τροπολογία 62. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 32 προ 4. Τροπολογία 20. Μπούσοι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 63. Μπουζόη, ζώει και Φόξ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 24 υπέρ κατά εγκρίνεται 25 υπέρ κατά εγκρίνεται 26 αποσύρθηκε 27 υπέρ κατά εγκρίνεται εκτιμώντας ήδη τροπολογία 28 Ζουβέν Βάις Γκέμπερ υπέρ κατά Ισχύει για όλο το κείμενο η αλλαγή της διατύπωσης. 29 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 30. Α, συγγνώμη, είναι 33, 33, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 34, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 35, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 36, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Εκτιμώντας 14. Κατά τμήματα ψηφοφορία, γιατί η κυρία Βάισμπεργκερ το ζήτησε, πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Όπω φαίνεται στον κατάλογο ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται 22 προς 14. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ωραία ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικός. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 33 ε, ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Μπουσόη. Uh, so we now move on to the second in this suite of... Uh, Πάμε τώρα στον κύριο Κορέα Δεκάμπος. Σύντομα, Πρόεδρε. Έχουμε κάνει μακροσκελή συζητήσει, συναντήσεις και χαίρομαι που τελικά καταλήξαμε σε σχεδόν πλήρη συμφωνία. Ευχαριστούμε. Ας αρχίσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Άρθρο 1, τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 12 καταπίπτει. 13. Ζουβέ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οι 15 και 16 καταπίπτουν. 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, σκέψεις. 1. Τροπολογία 1. Του εισηγητή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 11, μπουζόι. Ηλεκτρονικά να το δούμε αυτό για την 11. Open. The vote εγκρίνεται 24 προς 12. Τροπολογία 9. Βάις Γκέρμπερ Φόξ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2. Καταπίπτει. 10. Ζουβέν Βάις Γκέρμπερ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 9 δεν θα πρέπει να ψηφιστεί. Δεν θα πρέπει να είναι στον κατάλογο. Α, ναι. όντως, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Η 10 πέρασε. Τελευταία είναι η 3. Κορέα Δεκάμπου. Άρχεται η ψηφοφορία για την 3. The vote is open on Amendment 3 by, by the rapporteur. The vote is closed. Πέρασε Απορρίπτεται. 17 υπέρ, 19 κατά. Τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Uh, as everybody voted, the vote is closed. Uh, so that is carried by 34 in favour and 2 against. Περνάει η έκθεση 34 υπέρ, 2 ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια κύριε Κορέα Δεκάμπος. I think your first opinion, I think, for this Parliament. So the first of many, I'm sure. So thank you very much on Πάμε στην ε, έκθεση της κυρίας Ρούλε τώρα για τις δημόσιες προμήθειες. Κυρία Ρούλε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε, για να πάμε στην έκθεση του κυρίου Γκέξ. Να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και για, τις, ε, για την ε, διαθεσιμότητα που έδειξαν για συμβιβασμούς. Ε, κάποια ήταν αφιλεγόμενα σημεία, ειδικά οι, ε, δημόσια, οι συμβάσεις δημόσιου ιδιωτικού. Υπήρξαν κάποιε τροπολογίε, τι οποίε δεν μπορώ να υποστηρίξω, γιατί υπάρχει, υπάρχουν αποφάσει από το δικαστήριο που θα, αν, τις, αν ψηφίζαμε αυτέ τι τροπολογίε, θα έθεταν αναμφιβόλο πάλι αυτά που έχει συμφωνήσει και τελεσίδικα αποφασίσει το, το δικαστήριο. Δεν νομίζω ότι τώρα είναι η σωστή στιγμή να ζητούμε παραχωρήσει για τι επιχειρήσει μέσω μια οδηγία. Σε όλε τι συζητήσει που έκανα, σχεδόν κανένα δεν θέλει αυτή την οδηγία αυτή τη χρονική στιγμή. Και αν θα φαινόταν μέσω μιας αναθεώρησης ε, του συνόλου ε, των οδηγιών για τις ε, δημόσιες προμήθειες ότι υπάρχει ανάγκη, μόνο τότε θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε, αλλά όχι πιο πριν. Ευχαριστούμε για την δουλειά που έχετε κάνει. Οπότε ας αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Τίτλος, τροπολογία 18, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 20, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 19, υπέρ. Να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Vote open on amendment 19. Vote closed. Πέρας. 28 υπέρ, 8 κατά. Συμβαστική πρόταση 1. 21, οι 2 έως 27 τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 28. Ηλεκτρονικά. Α, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 προς 18. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 προ 21. 29. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Η 4 καταπίπτει. 56. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 2. Uh, the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 21 προς 14. Uh, so we now then move through to amendments 37 and 70. 57, 75 συγγνώμη, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Εγκρι... Εγκρίνεται. 41 αποσύρεται. Πάμε στην 38. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 39. Προσθήκη. Υπέρ. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 39. Uh, that is carried.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 40. Στήλερ. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Amendment 40. Vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 14 in favor, 20 against. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 49. Κρόιτσμαν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 53 και 54. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας Απορρίπτεται. 22 προς 11. 55. Κρότσμαν υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. της Επιτροπής περιφερειακή Ανάπτυξη. 6. Τροπολογία 6. Την ψηφίζουμε, την ψηφίζουμε. Α, καταπίπτει. Α, καταπίπτει, καταπίπτει. Πάμε στην 47. Ε, 57. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ, κατά. 59 υπέρ κατά απορρίπτεται όπως και 60. Πάμε στην παράγραφο 7. Υπέρ κατά απορρίπτεται. Φλόρενς υπέρ κατά απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 61 υπέρ κατά εγκρίνεται προσθήκη. Πάμε στην 66 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 9. Τροπολογία 73 Βερνιό. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 73 της κυρίας Βερνιό. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 26 προς 10. Πάμε στην ενοποιημένη τροπολογία από αρκετούς συναδέλφους. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. That is carried by 22. Εγκρίνεται 22 προς 14. Οπότε πάμε στην 71-74 που μπαίνουν στην ψηφοφορία ως προσθήκη. Ηλεκτρονικά να το δούμε. 71 και 74. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17 προς 15. 72 Κρόιτσμαν. Ε, προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. 72. Να το δούμε ηλεκτρονικά. Μπερδεύτηκε το ΕΛΚ. Τι έγινε. Θα το δείτε ότι θα απορριφθεί. Πέρας πληροφορίας. Ε, όπως σας είπα, 31 προς 4. Απορρίπτεται. Ο κύριος Κρόιτσμαν δυστυχώς δεν είναι η ώρα του ακόμα να επιβληθεί στην ομάδα μας, στην επιτροπή μας με τις τροπολογίες του. 77. Για την παράγραφο 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 84. Καταπίπτει. Πάμε στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. 5. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 11. Τροπολογία 82. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 83 της κυρίας ουρίουλε. Το κείμενο το έχετε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 84 της κυρίας Βάης Γκέρμπερ ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία της κυρίας Βάης Γκέρμπερ. The uh, vote is closed. Uh, that is carried by 23 votes to 13. Εγκρίνεται 23 προς 13. 85. Τροπολογία 85 και την παράγραφο 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 21 προς 15. 89. Υπέρ. 89. Άρχιδη ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 32 προς 3. 90. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 91. Σβάμπ. Υπέρ. Εγκρίνεται. 92. Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 95. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η καταπίπτει η Ρέτζι 8. 127 υπέρ. Εγκρίνεται. Διεθνές εμπόριο 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Διεθνές εμπόριο 8. Την κυρία Χάνσλικ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 129 καταπίπτει. Η 43 επίσης καταπίπτει. Πάμε στην παράγραφο 13. Τροπολογία 93. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 95 αποσύρεται. 94 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 98 καταπίπτει. Πάμε στην 102 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 101. Νομίζω θα την ψηφίσουμε ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία για την 101 του κυρίου Νικολέσκου. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 20 προς 15. 45 και 12. Να τα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Εγκρίνονται και οι δύο. 123. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, τι έγινε, μπερδευτήκατε. Ο κύριος Σφάπ χωρίς μικρόφωνο. Ψηφίζαμε τη 45 και τη 12, που είναι ταυτόσιμες, του κυρίου Πουπάκη. Είμαστε στην 123 τώρα. Λοιπόν, 123 πάλι. Υπέρ της 123. Κατά. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Παράγραφος 14. Συμβασική πρόταση 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στη 44. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15. 111. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 117. Υπέρ. Να τη δούμε ηλεκτρονικά αυτή. 117 του κυρίου Φαντεκάμπ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 προς 14. 118. Head. Α, αποσύρεται. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Αποσύρεται. Πάμε στην 113 της κυρίας Βερνιό. Άρχεται η ψηφοφορία για την 113. The vote is Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 21 προς 13. Θα ψηφίσουμε την 116. So, amendment 116 we vote as an addition. 116 την ψηφίζουμε ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. reject. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 προς 15. Ψηφίζουμε την 114 και την 115. Άρχεται η ψηφοφορία. 114-115. Uh, the vote is closed. Πέρας. Απορρίπτονται. 19 προς 14. Να είστε λίγο πιο γρήγοροι στις, ε, στην ψηφοφορία σας όμως όταν ψηφίζετε. 112. Άρχεται η ψηφοφορία για την 112. Vote Πέρας. Απορρίπτεται. 20 προς 16. 119. Νικουλέσκου. Προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 προς 13. Κρόιτσμαν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στην 97 και 99. 97 και 99. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. That's defeated. Πέρας. 21-15. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 11. Την 100 διορθώνει ο πρόεδρος. 100. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 21-15. 96. Βάις Κέρμπερ. Προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. 103 του κυρίου Τρενταφυλλίδη. 103. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται 23 προς 12. 24. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 προς 12. 126. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 122. Γκυγιόμ. De Jong. Άρχεται η ψηφορία για την 122 De Jong. De Vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 προς 14. Βερνιό, 128. Άρχεται η ψηφοφορία για την 128 της κυρίας Βερνιό. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 προς 14. Πάμε στις επόμενες τρεις που καταπίπτουν πάμε στην 130 υπέρ κατά εγκρίνεται 124 υπέρ κατά εγκρίνεται πάμε σε αρκετέ τροπολογίε να τι δούμε όλε μαζί από την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Όχι, όχι. Δύο. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Mr. Πέρας. Εγκρίνεται 18 προς 17. Τρία. Άρχεται η ψηφοφορία. Come on, Άντε συναδελφοί ψηφίστε. Κάντε λίγο γρήγορα γιατί παρατραβάει η ψηφοφορία. Πέρας. 22 προς 12 εγκρίνεται. 4. Βλάσεκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε σε μια σειρά τροπολογιών από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Χάνσλικ. Ένα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έντεκα, υπέρ κατά εγκρίνεται Τρία. Ηλεκτρονικά νομίζω να το δούμε. αρχιτή ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 προς 15. 4. αρχιτή ψηφοφορία για την 4. Uh, the vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται 18 προς 15. Είναι το 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5. Άρχεται η ψηφοφορία για την 5. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 προς 16. Είναι τα 6. Άρχεται η ψηφοφορία για την ίντα 6. Πέρας. Απορρίπτεται 19 προς 14. Είναι τα 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Είναι τα 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στα εκτιμώντας. 1, 2, 3, 4. Αποσύρονται. Πάμε στην 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά εγκρίνεται πάμε στα εκτιμώντας 7 Τη κυρία Βάιλερ άρχεται η ψηφοφορία The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται 20 προς 13. 17. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. Καλχάιν Φλόρενς. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία του κ. Φλόρενς. Πέρα, Εγκρίνεται 19 προς 16. Καταπίπτουν οι τροπολογίε του κ. Κρόιτσμαν. Πάμε στην 11 του κ. Κρόιτσμαν. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τα καταφέρατε κύριε Κρόιτσμαν. Τα καταφέρατε. Πέρασε η τροπολογία σας. 21 προς 13. Κύριος Δε, Άρχεται η ψηφοφορία για τη 12. Uh, the Πέρας. Απορρίπτεται. 22 προς 11. 15. Uh, uh Mr. 15. Uh, Υπέρ κατά εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. 40 De Jong 14 του κύριου Γιόγκ, συγγνώμη. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 προς 14. 16. Γιόγκ και 30 Τριανταφυλλίδης υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία για, το, για την γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφι, κα, ψήφος κατά. 28 in favour, no votes against, no abstentions. So thank you very much indeed to Heidi Ruler. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ρούλε, πολύ σημαντική έκθεσή της. Ευχαριστούμε και για την υποστήριξη που τους δώσατε. So, I think we have to... Ωραία. Να δούμε την έκθεση Γκρέσ. So, uh, Mr. Greg will speak at the στο τέλος θα πάρει το λόγο ο εισηγητής, ε, να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Και έχουμε και την ε, έκθεση του κυρίου Έγκστρομ, την οποία μπορεί να την ψηφίσουμε τα απόγευμα στην αρχή της συνεδρίας τελικά. Αλλά για την ώρα, ας περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Γκρέκ. Παράγραφος 1, τροπολογία 15 ρουσφόρ. Έναρξη ψηφοφορίας. Μήπως μπορείτε να ψηφίσετε λίγο πιο γρήγορα. Ένα κουμπάκι έχετε να πατήσετε. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 προς 12. 16. Ράπτη. Έναρξη ψηφοφορία για την τροπολογία 16. Πέρας. Εγκρίνεται 16 προς 14. Παρακαλώ να είστε γρήγοροι γιατί θα κλείνω γρήγορα τι ψηφοφορίε. Πατήστε γρήγορα το κουμπάκι σα. 17 τριανταφυλλίδη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 Ιβάνοβα παραγραφο 3. Κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται επίση. Του κυρίου Πουπάκη. Υπέρ. Τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Confirm. Τροπολογία 20. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Uh, the, vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται 22 προς 13. Τροπολογία 21. Τριανταφυλλίδης Δε Jong. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Κόμι. Έναρξη ψηφοφορίας. Uh, sorry, amendment 22. Thank you. Yes. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 προς 18. Τροπολογία 23 Ροσφόρ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 21 προς 13 ψήφι. Παράγραφος 6 Τροπολογία 29 φιλίδης. Υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Προφορική. Υπέρ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία του κυρίου Κρόιτσμαν. Πέρας. Εγκρίνεται. Ομοφωνία. Λίγο πιο γρήγορα το ΕΛΚ παρακαλώ. Αργούμε. Τροπολογία 25, Κρόιτσμαν. Έναρξη ψηφοφορία. Α, καταπίπτει. Oh, sorry, it was false. Okay. Right, okay. 24, sorry. Συγγνώμη, περνάμε στην 24. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Χαγνούγκ. Πρώτο τμήμα. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Λοιπόν, πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Uh, Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20, 20 προς 16. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα. Α, είναι της κυρίας Κόμη στη μέση. Ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τροπολογία 27 πρώτα. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρας. Άμαν, 18 όλα. Δεύτερο τμήμα. Χαγνόκ. Απορρίφθηκε η προηγούμενη. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Uh, the vote is ε, closed. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 προς 13. Παράγραφος 7. Τροπολογία 31 ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Ιβάνοβα. Έναρξη ψηφοφορίας. Compromise 4 was rejected. No. Yeah, that's right. So we, we, we then, yeah. It's all right. So the vote is open now. Έναρξη ψηφοφορίας. Uh, the vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Έναρξη ψηφοφορίας. Νομίζω θα απορριφθεί. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Όντως. Παράγραφος 8, τροπολογία 34, ροσφόρ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 35, κομφά, ως προσθήκη. Έναρξη ψηφοφορίας για την 35. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 19 προς 17. Καταπίπτει 33, πάμε στην 36 Κρόιτσμαν. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Άρα η 37 την ψηφίζουμε, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται του 20 ε, προς 15. 38 Ιβάνοβα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 23 προς 10. Τροπολογία 39 Φιλίδης, Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Παράγραφος 10, 41, τροπολογία Ροσφόρ. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία στη 42 της κυρίας Κόμη. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρα οι 42 και οι 40 καταπίπτουν. προφορική τροπολογία 47 έναρξη ψηφοφορία. ο συγγνώμη, χωρίς ηλεκτρονική ψηφοφορία, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 47 καταπίπτει, 46 έχει αποσυρθεί, 45. Χάντσλικ. α, κατα, καταπίπτει. Άρα φτάνουμε στο Κρόιτσμαν, 48. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 48, Κρόιτσμαν. 19 to 17. Πέρασε 19 έναντι 17. Και νομίζω ότι οι 43 και 44 καταπίπτουν. 49 που πάκης υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 50 ροσφόρ υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Προφορική 53 που εσύ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 53, η 53 καταπίπτει. Η 52, ψηφίζουμε την 52, με ονομαστική, με ηλεκτρονική. Closed. No, no, because you voted for the oral amendment. That, that is defeated. Απορρίπτεται. Για μία ψήφο. Α, η 53 κατέπεσε. Έχετε δίκιο. Παράγραφος 14. 57. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 τη 12. Η 55, 56, 54 καταπίπτουν. Παράγραφος 15. Προφορική του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα η 62 Α, α, έχει αποσυρθεί, εντάξει. Προτρέχεται. 63 Ψηφίζουμε την 63. Κατά. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66. 61. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 66. Κάρας. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 έναντι 14. 68 ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. So, 60, 68, 68 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 εναντί 16. 67. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 67. The vote is... Πέρας. 20 εναντί 13. 69. Ροσφόρ. Στην παράγραφο 17. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 71 γιατί 70 κατέπεσε υπέρ κατά εγκρίνεται. 72. Χάνσλεκ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 72. The vote is... Πέρας. 16 πέρα 17 κατά. 73. Κόμι. Υπέρ της τροπολογίας κατά εγκρίνεται. 74 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. Κανθά 76 αρχίζει η ψηφοφορία για την 76 πέρας απορρίπτεται 20 κατά, 15 υπέρ. Ε, συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρα 82 Λόκεγκάρτ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 82. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 έναντι 13. Παράγραφος 20. Jong Τριανταφυλλίδης υπέρ κατά απορρίπτεται. Ροσφόρ 84 προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 85 κάρας υπέρ κατά εγκρίνεται. 86 προφορική καμφέ αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται σοψηφία ψηφίζουμε την 86 υπέρ κατά άρα απορρίπτεται Lockegaard 87 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 88. Λόκεγκάρτ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Πέρασε και αυτή η τροπολογία συμβιβασμού. 4. Συμβιβασμού. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβασμού 5 υπέρ κατά επίσης εγκρίνεται. Άρα βρισκόμαστε στην παράγραφο 25 προφορική του κυρίου Τριανταφυλλίδη 107 αρχίζει η ψηφοφορία για την προφορική αυτή. Πέρας. Απορρίφθηκε 15 20, άρα ψηφίζουμε την 107 καθεαυτή υπέρ κατά Απορρίπτεται. 108 Τριανταφυλλίδη, Το κυρίου Τριανταφυλλίδη ξεχωριστή υπέρ κατά ε, απορρίπτεται. Και τώρα... Α, ε, καταπίπτει ολόκληρη και το δεύτερο τμήμα. Α, το ψηφίζουμε το δεύτερο. Δεύτερο τμήμα, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Αρχίζει η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Πέρασε. Εγκρίθηκε 17 έναντι 15. Κρόιτσμαν, παράγραφος 26, 112. Υπέρ, κατά. Απορρίφθηκε. 110, Χάνσλικ, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Χάθηκε 12 έναντι 23. Ροσφόρ 111 υπέρ κατά εγκρίνεται η 109 καταπίπτει 114 κάρας ε, τουν αρχίζει η ψηφοφορία για την 114 πέρας πέρασε 24 εναντί 10 113 προσθήκη Ροσφόρ αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας. Πέρασε 20 αντί 15. Τροπολογία 115. Ροσφόρ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 115. Ροσφόρ. Πέρας. Εγκρίθηκε 21 ψήφια έναντι 13. 116 έχει αποσυρθεί. Παράγραφος 28. Um, uh, paragraph, so amendment 120 καμφέν υπέρ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. 120 καμφέν. Closed. Πέρας. Εγκρίνεται 15 αντί 15. Ψηφίζουμε την 118 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 117 καταπίπτει, 119 προσθήκη, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 121. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 121. Uh, the vote is closed. Πέρας, εγκρίνεται. 24 εν 10, Χάντσλικ έχει αποσυρθεί, παράγραφος 29. 123 έως 126 υπέρ κατά εγκρίνεται 124 υπέρ κατά εγκρίνεται 125 αρχίζει η ψηφοφορία επί της 125 πέρας εγκρίνεται 19 έναντι 16 ψήφων 127 υπέρ κατά εγκρίνεται 128 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 129 αρχίζει η ψηφοφορία, επί της 129, πέρας, εγκρίθηκε 25, έναντι 10. 134 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 130 αποσύρεται και 131, 132. 132. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 133. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 135. 135. Υπέρ παρακαλώ. Κατά Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 137 αρχίζει η ψηφοφορία επί της 137. Uh, That is carried by... Πέρασε. Πέρασε. 138 138 αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίθηκε. 19 15. 139 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 14 ψήφων. 140 υπέρ κατά απορρίπτεται. 141. Ε, κάρας. Ε, ξεχωριστή ψηφοφορία ζήτησαν οι φιλελεύθεροι. Τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και αρχίζουμε τη ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. 141. Κάρας. Πέρας. Απερίφθη. 18. Κατά. 142 ράπτη υπέρ κατά σας παρακαλώ ε, ξανά 142 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απερίφθη για μία ψήφο 143 Ροσφόρ Λόκεγκάρτ υπέρ κατά Απορρίπτεται. 144. Κρόιτσμεν. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 144. Πέρας. Εγκρίθηκε 20 έναντι 13. 145 του Πρόεδρου. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 146 που πάκει υπέρ, κατά εγκρίνεται. 148 αποσύρεται και έχουμε μία προφορική, την 147 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 150, 30 φιλί. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 150. Πέρας. Απερίφθη. 20 κατά 14 υπέρ. 153 Χάντσλικ. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Μπορούμε να ε, ελέγξουμε. 153 Χάντσλικ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 3 υπέρ 29 κατά. Παρακαλώ να σηκώνει τα χέρια σαφέστερα. 151 κάρας τον αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is Πέρας. Εγκρίνεται. 21 15. 152 κατά καταπίπτει. 154 Κρόιτσμαν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 155 Ροσφόρ υπέρ κατά εγκρίνεται. 156 γκρέχ υπέρ κατά εγκρίνεται. 157 Λόκεγκάρτ προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 160 τουν Α, καταπίπτει, με συγχωρείτε. 158 κόμι. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 158. Πέρασε. Απερίφθη. 18 κατά. Έχουμε μία προφορική στην 159. Κάρας Ιβάνοβα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα 159 καταπίπτει. 166 ως προσθήκη. Αρχίζει η ψηφοφορία. 161 προσθήκη. Πέρασε εγκρίνεται. 19 έναντι 15. 161. 162 κάρα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 163 Χάνσλικ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Προφορική 164 Ράπτη υπέρ. Α, όχι, αρχίζει η ψηφοφορία επί της 164 Ράπτη. Πέρας εγκρίθηκε με 21 ψήφους εναντί 12. Άρα έχουμε Κρόιτσμαν ως προσθήκη, 165. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 23 εναντί 11. 166 κόμι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 167 κόμι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 168 30 Φιλίδης υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 171 Ροσφόρ. 171 ε, those in favor, those against. Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Άρα η 169. Α, όχι, με συγχωρείτε. Ψηφίζουμε την 169. 172 ε, αποσύρεται. 173. Α, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Άρα ψηφίζουμε την 174 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 175 υπέρ. Μάλλον, με συγχωρείτε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Περνάει 22 έναντι 12. Και τώρα, επειδή η επόμενη καταπίπτει, τι συμβαίνει λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτει και 178, 177 κόμι υπέρ, κατά. Περνάει. 179 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 181. Τριανταφυλλίδης de Γιόγκ. Αρχίζει η ψηφοφορία. 181. The vote is closed. Ε, απορρίπτεται. Ροσφόρ, 182 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 180. Κάρας Ιβάνοβα. Αρχίζει η ψηφοφορία. The closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 2014. 183 αρχίζει η ψηφοφορία. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λέει ο Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά εγκρίνεται συνεπώς 205 ξεχωριστή δική μου το πρώτο τμήμα λοιπόν της 205 υπέρ κατά εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται Άρα φτάνουμε στην 209. Κρόιτσμαν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Χάνσλικ. 210. Αρχίζει η ψυχοφορια Πέρας. Εγκρίνεται. 18 έναντι 16. 211 καταπίπτει, συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται και 221 τώρα, α με συγχωρείτε 222, αρχίζει η ψηφοφορία επί της 222, Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, όλες καταπίπτουν με συγχωρείτε. Προφορική 227 Ιβανόβα. Προφορική στη 227. Θα ήθελα να κάνω μία τροπολογία επί της τροπολογίας, δηλαδή στο readily available θα ήθελα να προσθέσουμε EU citizens. EU citizens των Ευρωπαίων πολιτών. Μία λέξη προσθέτουμε. Αν και είναι τελευταία στιγμή, μπορούμε να το δεχτούμε. Λοιπόν, ας δούμε τις προγενέστερες. all EU citizens. Μπορούμε να δεχτούμε αυτή την προφορική επί της προφορικής. Ψηφίζουμε την προφορική όπως ε, τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά εγκρίνεται. ...228 ράπτη υπέρ, αμάλλον ονομαστική. Για την προσθήκη 228 ράπτη αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 21 13. Άρα ας πάμε πίσω συνάδελφοι πάλι. Ψηφίσουμε τη 222. Γιατί κάναμε λάθος. Παράγραφος 58. 222. Αρχίζει η ψυχοφορία επί της 222. Πέρας. Απορρίφθηκε. Για μία ψήφο. 2-2-3 υπέρ κατά απορρίπτεται. 2-2-4 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται ισοψηφία. 225. Αρχι... Α, μάλλον ποιοι είναι υπέρ, λέει ο πρόεδρος, κατά επίσης απορρίπτεται και 226 αρχίζει η ψηφοφορία επί της 226 πέρας επίσης απορρίπτεται όλες απορρίπτονται σε αυτή τη σειρά 59α νέα 229 μπάστος ποιοι είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 2.30. Αρχίζει η ψηφοφορία. 230-233. Πέρας. Εγκρίθηκε. 19 16. Παράγραφος 60. Ροσφόρ. Αρχίζει η ψηφοφορία στη 231. Πέρας. Απορρίφθηκε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοφοριών. Θα ήθελα να, γίνει, να με βάλετε υπέρ. Είμαι υπέρ της τροπολογίας Κρόισμαν. Προστίκη λοιπόν. Uh, so, let's be clear. The rapporteur was against this, but is now in favor. No, no. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Mistake. it was a mistake. It was a mistake. It was a mistake. Okay, so 232, those in favor. 232. Those against. Κατά. Εγκρίνεται. 234 με μία προφορική καμφέ. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 234 προφορική. The vote is closed. Πέρας περναει 21 20-15. 235. Κρόιτσμαν υπέρ. Α, όχι, ονομαστική, αλλάζει ο πρόεδρος. Uh, the vote is closed. That's carried by 20 to 40. Πέρασε. 21-14. Ράπτη. 236. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ράπτη. Πέρασε 20 έναντι 13. Λοιπόν, αιτιολογικέ σκεψει 1. Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Πέρασε. 2. Γιόγκ Τριανταφυλλίδη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Περνάει 22 έναντι 13. Τρία, καμφέ, υπέρ κατά περνάει, εγκρίνεται Τέσσερα, κόμι υπέρ κατά αποχές περνάει Πέντε, γκρέχ υπέρ κατά εγκρίνεται Έξι, χαγνόκ υπέρ άμε συγχωρείτε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Περνάει. Η 7 καταπίπτει. 8 τριανταφυλλίδης. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα περνάμε στην 12. Κορέα Campos, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14. Μάλλον τελική ψηφοφορία επί της 14. Αρχίζει η ψηφοφορία στη 14. Κρόιτσμαν, Ροσφόρ. Πέρασε. Πέρασε 21 ψήφοι υπέρ, 13 κατά. Άρα ψηφίζουμε το κείμενο στο σύνολό του. Αρχίζει η ψηφοφορία επί του συνόλου, της έκθεσης δηλαδή. Πέρασε. Εγκρίνεται. 32-0. Τρεις αποχές. Συγχαρητήρια. να ολοκληρώσουμε. Έχουμε μια μικρή ψηφοφορία για την ε, ε, γνωμοδότηση του κυρίου Έγκστρομ, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε χωρίς διερμηνία. Παρακαλώ, ησυχία στην αίθουσα. Χωρίς διερμηνία, παρακαλώ. Ρωτάει ο πρόεδρος αν συμφωνεί.